Ε, λοιπόν, αρχίζει η συνεδρίαση της ακρόασής μας μαζί με την Επιτροπή Ελευθεριών, ΛΥΜΠΕ, με θέμα την κατάσταση των ε, εργαζομένων μεταναστριών σε αγροτικές περιοχές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, θα ήθελα να δώσω το λόγο στις βασικές μας ομιλήτριες η κυρία Φραντσέσκα Κομισάρη που είναι φωτογράφος από τη Σικελία και την έχουμε καλέσει από την Επιτροπή Γυναικών. <laughs> Ε, Καλημέρα σας. Μου δόθηκε δυνατότητα πριν από τέσσερα χρόνια να φτάσω στην Σικελία. Δεν κατάγομαι από τη Σικελία και για δυόμιση χρόνια ασχολήθηκα με το ζήτημα των γυναικών από τη Ρωμανία που εργάζονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της επαρχίας της Ραγκούσα στη Σικελία. Βλέπετε εδώ πέρα κάποιες από τις φωτογραφίες που έβγαλα την περίοδο αυτή. Βλέπετε εδώ πέρα μια θέα της κοιλάδας της Ραγκούσα τα τελευταία 30 χρόνια στην, εποχή, περιοχή αυτή τα πράγματα άλλαξαν πάρα πολύ. Από εκεί πέρα που καλλιεργόντουσαν κυρίως μικρά αγροτεμάχια και κυρίως αμπέλια, έχουμε πλέον όλο και περισσότερα θερμοκήπια. Και βλέπουμε ότι τελευταία χρόνια απασχολούνταν όλο και περισσότερο εργαζόμενοι από το Μαγκρέμπ, από τη Βόρεια Αφρική. Από τότε που εντάχθηκε η Ρουμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισαν να φτάνουν στην περιοχή εργαζόμενοι από την Ανατολική Ευρώπη και το τελευταίο διάστημα έχουμε δει πάρα πολλέ γυναίκε από τη Ρουμανία, οι οποίε απασχολούνται στα θερμοκήπια και τι γεωρικέ εκμεταλλεύσει τη Ραγκούσα. Οι γυναίκε αυτέ φτάνουν από μια συγκεκριμένη ζώνη τη Ρουμανία, την Μολδαβία, Σπακάο και Μποτοσάνη, από αυτέ τι βασικέ, τι δύο αυτέ περιοχέ, όπου ουσιαστικά η οικονομική κατάσταση είναι πάρα πολύ δεινή. Με το ζόρι τα βγάζουν πέρα, φτάνουν λοιπόν στη Σικελία προκειμένου να καταφέρουν να έχουν έναν ελάχιστο μισθό, μια ελάχιστη αμοιβή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν φτάνουν στην Ιταλία, φτάνουν στη ζώνη αυτή της επαρχίας της Ραγκούσα και λαμβάνουν μισθούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαμηλοί αλλά σαφώς πάρα πολύ ψηλότεροι από αυτούς που θα λάμβαναν στη Ρουμανία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τη θέση των γυναικών αυτών σε αυτή την ε, περιοχή, γιατί πραγματικά τροποποιείται με την παρουσία τους ε, η πολιτισμική και γεωργική ε, εικόνα της περιοχής αυτής. Οι γυναίκες αυτές κερδίζουν πολύ λιγότερα χρήματα, λαμβάνουν πολύ χαμηλότερους μισθούς από ότι οι μετανάστες από τις χώρες του Μαγκρέμπ στο παρελθόν είχαν καταφέρει μέσω συνδικαλιστικών οργανώσεων να καταφέρουν να έχουν οι προερχόμενοι από τι χώρε του Μαγκρέπ εργαζόμενοι πάνω κάτω τους ίδιου μισθού με του Ιταλού. Αυτή τη στιγμή οι γυναίκε από τη Ρουμανία κερδίζουν το πολύ 10 με 20 ευρώ την ημέρα μόνο απασχολούνται κυρίως γυναίκες και αυτό ταράζει εντελώς το υφιστάμενο οικονομικό σύστημα της περιοχής. Παλαιότερα γυναίκες δεν εργάζονταν στον γεωργικό τομέα στην περιοχή. Οι γυναίκες αυτές φτάνουν συνήθως με την οικογένειά τους, δηλαδή με μικρά παιδιά, πολλές φορές φτάνουν και μόνες τους, πολλές φορές μένουν και μόνες τους ε, όσο διάστημα παραμείνουν στην Σικελία τα δύο αυτά δύο-δυόμιση χρόνια που εργάστηκα στην περιοχή αυτή, στα πλαίσια αυτού του φωτορεπορτάζ, συνειδητοποίησα ότι το όλο κύκλωμα πλέον απασχόλησή του είναι πάρα πολύ κλειστό. Τα άτομα αυτά φτάνουν με πούλμαν από τη Ρουμανία, φτάνουν στον σταθμό της Βιτόρια, που είναι η βασική πόλη της επαρχίας της Ραγκούσα, όπου γίνονται αυτές οι προσλήψεις αναλαμβάνονται άμεσα από άλλους Ρωμάνους εργαζόμενους που βρίσκονται ήδη στην περιοχή και τις μεταφέρουν άμεσα στα θερμοκήπια αυτά που μένουν πραγματικά κλεισμένες εκεί. Πρόκειται για γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες είναι μικρές. Ε, αναφερόμαστε εδώ πέρα σε επιχειρήσεις που απασχολούν τρει-πέντε βασικού εργαζόμενου. Είναι ουσιαστικά οικογενειακέ γεωργικέ επιχειρήσει μικρή κλίμακα. Τώρα, στα θερμοκήπια αυτά που εργάζονται οι γυναίκες αυτές, όχι μόνο εργάζονται, αλλά ζουν και εκεί και πρέπει να αντιμετωπίσουν ε, πάρα πολλές άλλε δαπάνες. Καλούνται πολλές φορές να πληρώσουν ακόμα και τη διαμονή τους, ενώ διαμένουν μέσα στα θερμοκήπια ουσιαστικά πολλές φορές ζούνε σε αποθήκες, γεωργικές αποθήκες, εκεί, εκεί που λογικά έχουμε τα φυτοφάρμακα, τα χημικά προϊόντα, τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στην ε, γεωργία. Καλούνται λοιπόν να διαμορφώσουν τους χώρους αυτούς ε, και να τους καταστήσουν ε, σπίτια, αν μπορούμε ποτέ να αποκαλέσουμε σπίτια τις αποθήκες αυτές. Πολλές φορές δεν έχουν ηλεκτρικό, άλλες φορές δεν έχουν τρεχούμενο νερό. Το χειμώνα κάνει πάρα πολύ κρύο και στις ε, ψευτοκατοικίες ουσιαστικά αυτές ε, οι γυναίκες ε, διαβιούν πάρα πολύ κοντά στις, στα θερμοκήπια. Το βλέπετε και αυτό σε αυτή τη φωτογραφία, όπου το σπίτι αυτό, η αποθήκη, βρίσκεται πραγματικά πολύ κοντά στα θερμοκήπια. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λοιπόν, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Είναι συνεχώς σε επαφή με διάφορα χημικά προϊόντα. Πάρα πολλές γυναίκες καταλήγουν στο νοσοκομείο, στο μοναδικό νοσοκομείο που έχει η περιοχή αυτή με πάρα πολλά συμπτώματα τα οποία έχουν να κάνουν ε, με την ε, εγκύτητα αυτή που υπάρχει με τα χημικά προϊόντα. Έχουν δραματικά προβλήματα, έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ακριβώς επειδή βρίσκονται συνεχώς σε επαφή με τις ουσίες αυτές, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εργασίας, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πολλές από τις γυναίκες αυτές ε, κατοικούν λοιπόν σε αυτά τα παραπήγματα, καλούνται να αναλάβουν τις ίδιες ε, εργασιακές ευθύνες με τους άντρες, δουλεύουν τις ίδιες ώρες με τους άντρες και οι γυναίκες αυτές αναγκάζονται να πάρουν μαζί τους και τα παιδιά τους. Ορισμένες ε, αφήνουν τα παιδιά τους και στην Ρουμανία σε άλλους συγγενείς και προσπαθούν να τους στέλνουν τακτικά χρήματα. Πάντως, εν γέννη υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην περιοχή αυτή, παιδιά που έχουν έρθει μαζί με τις μητέρες τους οι οποίες ε, εργάζονται στα θερμοκήπια, παιδιά τα οποία δεν πηγαίνουν προφανώς στο σχολείο, δεν έχουν καταφέρουν να έχουν πρόσβαση οι γυναίκε αυτέ στο εκπαιδευτικό σύστημα, αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την μη γνώση τη ταλική γλώσσα. Δεν γνωρίζουν επίση πώ λειτουργεί το Ιταλικό σύστημα, όχι μόνο το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά εν γέννη το ταλικό σύστημα. Και το βασικό πρόβλημα που έχουν οι γυναίκες αυτές είναι η απομόνωσή τους. Μια απομόνωση που έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχουν μέσα μεταφοράς, δεν υπάρχουν δημόσια μέσα μεταφοράς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις γυναίκες αυτές να φύγουν τουλάχιστον από την περιοχή αυτή των γεωρικών εκμεταλλεύσεων και να πάνε προς γειτονικές πόλεις και χωριά. Καταλαβαίνετε ότι ε, όταν οι γυναίκες αυτές πληρώνται σε καθημερινή βάση 10 με 20 το πολύ ευρώ και ένα ταξί κοστίζει τουλάχιστον 25 ευρώ για να τους πάει στην πιο γειτονική πόλη, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορούν ποτέ να πάρουν κάποιο ταξί για να φύγουν από αυτή την περιοχή. Οι γυναίκες αυτές ε, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Ε, πολλές φορές χρειάζεται να κάνουν διάφορες χάρες στους εργοδότες τους προκειμένου να καταφέρουν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, προκειμένου να καταφέρουν απλώς να βρουν κάποιον που θα τους βοηθήσει να πάνε σε μια γειτονική πόλη χωριό. Βλέπετε εδώ πέρα την περίπτωση μιας γυναίκας η οποία ζει μαζί με τα παιδιά της στην περιοχή αυτή. Βλέπετε ένα από τα παιδιά εδώ πέρα. Το βράδυ κλείνουν πραγματικά τις πόρτες, τους φράκτες όλων αυτών των θερμοκηπίων προκειμένου να μην καταφέρουν να πάνε πουθενά. Το παιδί αυτό δεν έχει καταφέρει να πάει σε σχολείο. Ευτυχώ υπάρχει μία μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με την εμπορία ανθρώπων και που βοηθά τους ανθρώπους αυτούς. Το παιδί αυτό και η οικογένειά του έχει πάρα πολλά προβλήματα, δεν μιλάνε την Ιταλική γλώσσα, αλλά δεν καταφέρουν καν να βγουν από το χώρο αυτό της ε, γεωρικής εκμετάλλευσης, έχουν πάρα πολλά προβλήματα διατροφικά τρώνε ουσιαστικά μόνο πολέντα και ένα κομμάτι τυρί. Καταλαβαίνετε ότι στο τέλος της εβδομάδας ο συχνός αυτός μισθός που λαμβάνουν δεν τους επιτρέπει να αγοράσουν κάτι άλλο και το τυρί αυτό που τους δίνουν στο τέλος της εβδομάδας είναι ένα δώρο εντό αγωγικών που τους δίνει ο εργοδότης πέρα από το μισθό τους. Επίσης, τα παιδιά και οι γυναίκες πέφτουν ε, θύματα εκμετάλλευσης, κακοποίησης, όχι αναγκαστικά από τους εργοδότες αλλά και από τους υπόλοιπους διαμένοντες ενήλικες στην ε, γεωργική αυτή εκμετάλλευση. Τα παιδιά αυτά, καθότι οι γονείς τους εργάζονται 12 και πάνω από 12 ώρες ε, κάθε μέρα στη γεωργική εκμετάλλευση, πολλές φορές πέφτουν θύματα εκφοβισμού από άλλα παιδιά ή άλλους ενήλικους που βρίσκονται στην περιοχή. Η κακοποίηση αυτή και η εκμετάλλευση βέβαια δεν αφορά μόνο τα παιδιά αλλά και τους ίδιους ενήλικέ. Θα ήθελα να φερθώ εδώ πέρα στην περίπτωση της Νικολέτας, μία από τις ελάχιστε γυναίκες που φάσει να καταγγείλει τα φαινόμενα κακοποίηση και εκμετάλλευσης. Το πρόβλημα είναι ότι είναι ελάχιστε οι καταγγελίε γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποια ανταπόκριση. Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή α, ένα συγκεκριμένο σύστημα που θα μπορούσε να υποστηρίξει τι γυναίκε αυτέ. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εργοδότε οι οποίοι υποδέχονται τόσο εγωικών τι γυναίκε αυτέ θέτοντα ένα όπλο δίπλα στον κρόταφό του ουσιαστικά αναγκάζοντάς τους να αποδεχθούν πάρα πολλές συνθήκες οι οποίες θα ήταν απαράδεκτες σε άλλες χώρες. Είναι λοιπόν μία από τις λίγες γυναίκες στην Νικολέτα που φάσισε να καταγγείλει την κατάσταση αυτή. Όταν ήταν ε, έγκυος το τέταρτο παιδί της, την απείλησε ο εργοδότης της ότι θα την απειλούσε, ότι θα την απέλει, με αν δεν του πρόσφερε διάφορες σεξουαλικές χάρες και μάλιστα ακόμα και ο ίδιος ο σύζυγός της την πίεζε να ενδώσει στον εργοδότη προκειμένου να μην χάσει τη δουλειά της. Αποφάσισε λοιπόν δεν μπορούσε να ανοιχτεί πλέον την κατάσταση αυτή και ε, κατήγγειλε τον εργοδότη. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη μόνο γυναίκα που έχει κάνει κάτι τέτοιο από όλε αυτέ τι γυναίκε που εργάζονται στην περιοχή και οι οποίε έχουν πέσει θύμα κακοποίηση και εκμετάλλευση. Οι περισσότερες γυναίκες ζουν σε τέτοια ε, παραπήγματα, βοηθητικά κτίσματα, τα οποία υπάρχουν δίπλα στις ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αναγκάζονται να αφήνουν ανοιχτές τις πόρτες, βρίσκονται κατά αυτόν τον τρόπο από τη συνεχή επιτήρηση των εργοδοτών και οι περισσότερες από τις γυναίκες αυτές είναι ή αισθάνονται θύματα. Παρ' όλα αυτά δεν το παραδέχονται αυτό γιατί έρχονται ουσιαστικά από παρόμοιες καταστάσεις ε, στην χώρα τους και ο βασικός τους ε, στόχος είναι να καταφέρουν να εργαστούν, να διατηρήσουν την εργασία τους για να στείλουν χρήματα πίσω στο σπίτι τους ε, για να καταφέρουν εκεί πέρα να συντηρήσουν γονείς, συγγενείς και παιδιά. Οι περισσότερες λοιπόν από αυτές αποδέχονται και υπομένουν σιωπηλά καταστάσεις εξευτελιστικές. Έχουμε λοιπόν εργαζόμενες ε, γυναίκες ε, οι οποίες ε, υφίστανται απαράδεκτες συνθήκες. Ουσιαστικά υπάρχουν διάφορε μη κυβερνητικέ οργανώσει που αντιμετωπίζουν τι γυναίκε αυτέ σαν να ήταν άστεγες γυναίκε, ενώ στην πραγματικότητα είναι γυναίκε που απασχολούνται επί τόπου, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε και αυτέ να έχουν τι συνθήκε που προβλέπονται στι συλλογικέ συμβάσει, τι συνθήκε που προβλέπονται για του υπόλοιπου Ιταλούς. Προφανώ όμω δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πράξη. Πολλέ από τι γυναίκε αυτέ αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ιταλία και δεν αντέχουν άλλω συνθήκε αυτέ. Επιστρέφουν στη Ρουμανία, αλλά μετά από λίγο αποφασίζουν να γυρίσουν στην Ιταλία για να εργαστούν πάλι στα θερμοκήπια. Ακριβώς επειδή όταν γυρίσουν στη Ρουμανία ε, μένουν χωρίς δουλειά εκεί, δεν έχουν τα παρέτα μέσα για να τα βγάλουν πέρα, οπότε παρά τη, θε... παρά θέλησή τους επιστρέφουν στη Σικελία. Επίσης, ε, πολλές από τις ε, γυναίκες αυτές γνωρίζουν ότι ε, δεν έχουν κάποια εναλλακτική, ότι προκειμένου να μείνουν άνεργες στην ε, Ρουμανία προτιμούν να επιστρέψουν στην Ιταλία αποδεχόμενες συνθήκες αυτές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κομισάρη. Θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Τράγκητσα, Γενική Γραμματέα ε, της Εθνικής Υπηρεσίας Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών από τη Ρουμανία αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ε, Γυναικών ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να σας απευθύνω το λόγο. Επίσης, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για αυτά τα θέματα. Για τη ρουμανική κυβέρνηση, πρόθεση των ίσων ευκαιριών ε, μεταξύ και γυναικών, η προστασία των κοριτσιών και των γυναικών στη χώρα μας, αλλά και εκτός των συνόρων μας, είναι βασικά στοιχεία και θεμελιώδεις αρχές μιας κοινωνικής δημοκρατίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά ε, τα θέματα αυτά και συγκεκριμένα αυτό που μας απασχολεί σήμερα η μετανάστευση. Ε, ε, η σημερινή ρουμανική κυβέρνηση που ψηφίστηκε από τη Ρουμανική Βουλή, έχει κάνει πρόταση νόμου για το σεβασμό των γυναικών, της κατάστασης των γυναικών και την προστασία τους. Εξού και ο δικός μας οργανισμός, τον οποίο σήμερα εδώ εκπροσωπώ. Τι γίνεται με τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αγροτικές περιοχές και εκμεταλλεύσεις. Έχουμε μεγάλο εργατικό δυναμικό και νεαρό εργατικό δυναμικό ε, που εργάζεται στο εξωτερικό. Συνεργαζόμαστε με διάφορους οργανισμούς ε, για ε, να βοηθούν, για να προστατεύονται οι Ρουμάνοι από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, κακοποίηση και άλλες. Είναι από τις βασικές χώρες που προμηθεύει χέρια η Ρουμανία σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχουν πάρα πολλέ μεταναστευτικέ ροέ εσωτερικής μετανάστευση. Δύο εκατομμύρια είναι οι Ρουμάνοι που εργάζονται στο εξωτερικό και από τα δύο εκατομμύρια το 47% είναι γυναίκες. Οι γυναίκες λοιπόν μετανάστριε γνωρίζουν πολλούς κινδύνους ε, τους οποίους δεν ήξεραν στο παρελθόν και δεν θεωρούν ότι προστατεύονται ε, στην αγορά εργασίας. Ε, υπάρχουν εκθέσεις που τεκμηριώνουν ε, τους ε, κινδύνους που αντιμετωπίζουν για κακοποίηση, εκμετάλλευση, ακόμα και τράφικινγκ, διακίνηση. λοιπόν, είναι πάρα πολλές οι κακοποιήσεις και οι καταχρήσεις. Η Ρουμανική Διασπορά είναι πάρα πολύ ε, στο εξωτερικό. Οι γυναίκες όμως κινδυνεύουν ιδιαίτερα γιατί δεν έχουν ε, νομική προστασία και πολλές φορές ε, πέφτουν θύματα δουλεμπόρων και διακινητών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Ένα υποσύνολο ε, αυτών είναι ε, οι μετανάστρες που εργάζονται σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Πολλές φορές πρόκειται για σύγχρονες ε, μορφές δουλείας. Είναι μια εργασία χωρίς νομική προστασία, με συνεννόηση ή συνενοχή ενός Ρουμάνου ενδιαμέσου Ε, ενώ στις χώρες όπου υπάρχουν πολύ περισσότερες Ρουμάνες όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία υπάρχει και συνεργασία διπλωματική της δικής μας κυβέρνησης με τις πρεσβείες. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει προστασία ε, σε τοπικό επίπεδο από τις κυβερνήσεις δηλαδή των χωρών αυτών για να αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις και να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των δικών μας πολιτών που εκτίθενται σε κίνδυνο. Έτσι λοιπόν, η ρουμανική κυβέρνηση ε, εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή με τρόπο διαφρομένο, συνεπή και συνεκτικό και έχει λανσάρει μια εθνική καμπάνια για την ενημέρωση των πολιτών για την κατάσταση που επικρατεί ανά τον κόσμο ε, σε συνεργασία με τα διάφορα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και με άλλους οργανισμούς και θεσμούς έτσι ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους οι Ρουμάνες εργαζόμενες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θέλουμε να στηρίξουμε και τους Ρουμάνους που επαναπατρίζονται. Το Υπουργείο Εργασίας έχει ε, προβλέψει διάφορους μηχανισμούς ενημέρωσης και προστασίας για τους Ρουμάνους πολίτες που ε, ζουν και εργάζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και μάλιστα ως οδηγός του Ρουμάνου εργαζομένου που έχει εγκριθεί και ισχύει σε 21 χώρες αναφέρεται σε 21 χώρες και στο δίκτυο Γιούρες. Έχουμε και έναν οδηγό επίσης για τις συνθήκες εργασίας, τα δικαιώματα που έχουν τα μέλη της οικογένειας, το δικαίωμα ε, στη κοινωνική ασφάλιση, στα επιδόματα ε, ανεργίας, ε, και άλλα. Επίσης ενημερώνουμε τους πολίτες για τους κινδύνους που υπάρχουν ε, δωρεάν αν το επιθυμούν και για τις ε, διάφορες δομές ε, διαμεσολάβησης. Είναι 45 οι συμβουλοί του Γιούρες που βοηθούν τους πολίτες σε διάφορες περιοχές της Ρουμανίας. Έχουμε επίσης εργαζομένους 35 τον αριθμό που έχουν ως αντικείμενο εργασίας τους την προστασία των Ρουμάνων εργαζομένων στο εξωτερικό ε, αναγεωγραφική περιοχή. Για όσους επιθυμούν να επιστρέψουν, ε, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενημερώνουν και βοηθούν τους ε, επαναπατριζομένους για την πρόσβαση στην εργασία, τη διαμεσολάβηση, τον επαγγελματικό βίο και επίσης συμβουλές για την έναρξη επαγγέλματος ή την ίδρυση επιχείρησης ε, και αναγνώριση των προσόντων που έχει κάποιος αποκτήσει και των δεξιοτήτων εκτός της επίσημης εκπαίδευσης. Και με τις γυναίκες που εργάζονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχουμε στήριξη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε η γεωργία να είναι ένας κλάδος πιο ελκυστικός και για τα δύο φύλλα. Υπάρχει εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξη της υπαίθρου 2014-2020 με ε, μέτρα που συνάδουν με το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο των ε, κρατών μελών. Έτσι, όλοι οι αρμόδιοι θεσμοί για την πρόθεση της ισότητας ανδρών και γυναικών συμμετέχουν με παρακολούθηση από τα αρμόδια Υπουργεία και έτσι επιμορφώνονται ζευγάρια για την καταπολέμηση ε, των διακρίσεων ε, και με άλλα προγράμματα, με ΣΔΙΤ, από το πρόγραμμα LEADER, έχουμε χρησιμοποιήσει κάποια κριτήρια επιλογής, επιλεξιμότητας και λαμβάνουμε υπόψη και τη διάσταση του φύλου για να μην γίνονται διακρίσεις. Το ίδιο πρόγραμμα βοήθησε έμεσα ή άμεσα για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για γυναίκες ή να βελτιωθούν οι υφιστάμενες. Έτσι αυξάνεται και η παραγωγικότητα και η οικονομική ε, ανάπτυξη ε, με προώθηση της ισότητας των φύλων και ε, άρση των διακρίσεων. Επίσης, ενισχύουμε και τις δομές στην Ήπεθρο, την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την μετακπαίδευση μετά το σχολείο, ακόμα και τα νηπιαγωγεία για να μην υπάρχουν διακρίσεις στην πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ε, και στην Ήπεθρο ε, βελτιώνουμε την εκπαίδευση για να υπάρχουν και περισσότερες ευκαιρίες. Στη Ρουμανία λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει βούληση ε, να γίνουν όλα αυτά κτήμα των γυναικών και να υλοποιηθεί και ε, στη Ρουμανία η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2016-2019 για την ισότητα των φύλων. Κάνουμε διάφορες ε, ενέργειες επίσης για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας συνοδεύεται από ειδικά μέτρα. Θέλουμε να μεταφέρουμε στην πράξη και να υλοποιούμε τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αρθεί κάθε είδους διάκριση κατά των γυναικών. Υπάρχουν κάποιες συστάσεις επίσης για τη Ρουμανία. Ξέρετε ότι η Ρουμανία έχει κυρώσει ε, τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ε, που είναι σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της ενδοοικονικής. Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία, με την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό, την κυρία Βιωρίκα Νταντσίλα, ε, θέλει να αλλάξει τα πρότυπα και τα στερεότυπα για τις γυναίκες στη Ρουμανία. Αν μου επιτρέπετε να φέρω δύο νομοθετικές προτάσεις. Το νομοσχέδιο για την ισότητα ε, ευκαιριών και τη ρύθμιση κάποιων επαγγελμάτων όπως είναι το επάγγελμα του εμπειρογνώμονα έτσι ώστε να μην εμποδίζονται οι γυναίκες ε, στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Και το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής ε, βίας ε, σύμφωνα με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Εκεί έχουμε βάσει της σύμβαση αυτής και ενός άρθρου πρόταση για ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας με ειδικέ ε, ρήτρε και εντολές προστασίας και απαγόρευσης ε, προσέγγισης. Τώρα έρχομαι στο θέμα που μας απασχολεί σήμερα. Αυτό το θέμα με τις Ρουμάνες εργαζόμενες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό και άλλη μια ευκαιρία για την κυβέρνησή μας να διατρανώσει πόσο σημαντική θεωρεί την πρόθεση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, η Βερίκα Ταντσίλα είναι πρωθυπουργό της χώρα σα και εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και στην Επιτροπή μα ε, ήταν πολύ δραστήρια ευρωβουλευτή. Είναι πραγματικά ε, πολύ θετικό το γεγονός ότι ακούσαμε όλα αυτά τα στοιχεία για τη στρατηγική που έχετε χαράξει στη χώρα σας. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Λοιπόν, το, ο λόγος τώρα στην κυρία Σόρταλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ως τελευταία ομιλήτρια θα έχω την ευκαιρία βεβαίω να αναφερθώ σε κάποια θέματα τα οποία έχουν ήδη ακουστεί. Πρωτού όμω πω οτιδήποτε, ε, οτιδήποτε για τις ε, μετανάστριες εργαζόμενες, θα ήθελα να πω κάτι για, για την γενική κατάσταση της γεωργίας στην Ευρώπη. Η γεωργία εξακολουθεί να είναι ο χώρος, ο τομέα στον οποίο υπάρχουν μεγαλύτερε έμφυλε ανισότητε. Πολύ, πολύ σπάνια οι γυναίκε κληρονομούν ε, γη, ε, και αποτελούν ιδιοκτήτες της γης. Αυτό είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στην, ε, στην βόρεια ε, ε, Ευρώπη. 16% μόλις στο Ηνωμένο Βασιλείο. Και αυτές οι γυναίκες συνήθως είναι γυναίκες που έχουν κληρονομήσει τη γη από τον άντρα τους που πέθανε και το κρατούν για τους γιους τους. Ε, το, το ίδιο ισχύει και στην Νορβηγία και στην ε, Ιρλανδία. Στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ε, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Εκεί υπάρχουν περισσότερες γυναίκες ιδιοκτήτριες γης. Ε, οι, ε, οι εργαζόμενες λοιπόν στη Γεωργία αποτελούν τις μεγαλύτερες, αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ανισότητες από την άποψη του, του φύλου. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση όπου ε, οι γυναίκες ε, αντιμετωπίζουν παρενόχληση, διακρίσεις και υπάρχει μάλιστα και μια αιτιολόγηση αυτών των συμπεριφερών ε, στην Γεωργία. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτό κατά νου, ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες από άποψη φύλου. Άρα είναι, είναι σαφές ότι οι περισσότερες μετανάστες γυναίκες που εργάζονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις εργάζονται για ε, Εδώ βλέπετε ε, μια φωτογραφία από το Φέρμο Μάρτ. Τη δείχνω αυτή τη φωτογραφία γιατί υπάρχει μόνο μία γυναίκα σε ολόκληρη την αίθουσα αυτή. Ε, θέλω να μιλήσω για γυναίκες που μετακινούνται και εργάζονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις εντός Ευρώπης. Εγώ έχω ζήσει τα τελευταία 20 χρόνια στη Βόρεια Ιρλανδία. Θέλω να σας μιλήσω λοιπόν για το τι συμβαίνει στον τομέα της μεταποίησης τροφίμων εκεί ε, αλλά και για το τι συμβαίνει στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις καλλιέργειας μανιταριών κυρίως. Πριν από λίγο καιρό ήταν ανάγκη να εξηγηγούμε σε όλους που είναι ακριβώς η Βόρεια Ιρλανδία. Πλέον νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους στην Ευρώπη ποια, ποια είναι η Βόρεια Ιρλανδία. Βλέπετε εδώ είναι το βόρειο κομμάτι της νήσου της Ιρλανδίας, αλλά είναι κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου. Λοιπόν, Έχοντας εξετάσει λοιπόν την έκθεση αυτή, ε, τονίζεται εκεί και η μη διαθεσιμότητα στοιχείων για τις γυναίκες αγρότησες μετανάστες. Υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία για το τι ακριβώς συμβαίνει. Γνωρίζουμε ότι ε, περισσότεροι άνδρες εργάζονται στις γεωργικές δουλειές, αλλά και αυτό ε, ποικίλει ανάλογα με τον ε, κλάδο και τον τομέα. Ε, συνήθως οι γυναίκες προσλαμβάνονται σε συγκεκριμένου κλάδους, φράουλες για παράδειγμα στην ε, Ισπανία, γιατί θεωρούνται ε, πιο κατάλληλες λόγω των λεπτών χεριών που έχουν. Ταυτόχρονα ε, πολλές φορές προσλαμβάνονται μαζί με τα, παιδιά τους για να είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψουν και στην, στις αιστείες τους, στις πατρίδες τους μετά το τέλος της σεζόν της καλλιεργητικής περίοδου είναι χαμηλά αμοιβόμενες αυτές οι δουλειές. Είναι δουλειές όπου συμπιέζονται οι μισθοί και οι αμοιβέ είναι πολύ σκληρή δουλειά, είναι εποχιακή η δουλειά αυτή και κάποιες φορές αναφέρεται ότι πολλές από αυτές τις δουλειές θα μπορούσαν και να αυτοματοποιηθούν και να γίνονται από μηχανές, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει τόσο φτηνό εργατικό δυναμικό διαθέσιμο, δεν υπάρχουν και κίνητρα ε, ώστε να αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία. Αν, λοιπόν, αν και λοιπόν οι, ε, εργαζόμενοι αυτοί τυπικά ε, είναι νόμιμοι, λαμβάνουν πάρα, πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς σε πάρα πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, συνθήκες. Από τις έρευνες λοιπόν ε, που έχω διαβάσει, την έκθεση Πότερ και Χάμιλτον, αλλά και από τη δική μου δουλειά, ε, προκύπτει ότι υπάρχει ένας τεράστιος βαθμός φόβου. Οι άνθρωποι πραγματικά φοβούνται, δεν ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους, δεν, δεν, ε, πολλές φορές προσλαμβάνονται μέσα από γραφεία από πρακτορία ε, τα οποία τους φέρουν στην άλλη χώρα. Δεν ξέρουν για ποιον ακριβώς δουλεύουν. Δουλεύουν για τον αγρότη, για τον γεωργό, δουλεύουν για το, για το πρακτορείο αυτό. Δεν ξέρουν τίποτα για, τις, ε, για τα δικαιώματά τους και αυτό προκαλεί έναν φόβο ο οποίος είναι έκδηλος. Υπάρχουν διάφορα μειονεκτήματα βεβαίως για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτές τις γυναίκες, και αδυναμία, ε, ε, ε, ελλείψεις ως προς την γνώση της γλώσσας, δεν γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει σε σχέση με τους σπιτονικοκύριδες τους, που πολλές φορές τους παρέχουν ε, ακατάλληλα καταλήματα ε, και πολλές φορές δεν, ε, δεν, δεν υπάρχουν ούτε καν δυνατότητες μεταφοράς τους, μεταφέρουν οι ίδιοι οι εργοδότες τους. Αυτό βεβαίως προκαλεί μια φοβερή απομόνωση αυτών των, των γυναικών από την, από την υπόλοιπη κοινωνία. Επίσης υπάρχουν σοβαρά στοιχεία που μας δείχνουν ότι δεν πληρώνονται οι ε, δεν ενημερώνονται οι εργαζόμενες αυτές για το ποια είναι τα δικαιώματα Και θέλω να πω τώρα κάτι συγκεκριμένα για, τον, για τις γυναίκες που εργάζονται στον τομέα μεταποίησης τροφίμων. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η σημερινή μας εκδήλωση δεν αφορά μόνο γενικά τις γυναίκες σε ιερουργικές εκμεταλλές αλλά και τις γυναίκες σε αγροτικές περιοχές εν γέννη γιατί υπάρχουν και πολλές γυναίκες που ε, εργάζονται όχι μόνο στα χωράφια αλλά και στα εργοστάσια μεταποίησης τροφίμων και σε αυτόν τον τομέα συγκεκριμένα ε, εγώ έκανα έρευνα στη Βόρεια Ιρλανδία και διαπίστωσα ότι υπάρχουν πάρα, πολλές, κατηγορίες ξένων μεταναστριών. Υπάρχουν ε, Ρουμάνες, Ουκρανές, Πορτογαλίδες, Λιθουανές, ε, Λετονές. Και εκεί οι γυναίκες αυτές αναφέρουν συστηματικά πόσο υποαμείβονται, πώς πάντοτε οι επιστάτες είναι άντρες πως ε, ε, ε, δεν πληρώνονται υπερορίες, πολλοί, πολλές εργαζόμενες έρχονται από την, προέρχονται, κατάγονται από την Λετωνία και πολλές φορές ακολουθούν άλλους, άλλες συμπατριώτησές τους που έχουν πάει στην, στην εκάστοτε χώρα ε, νωρίτερα αντίθετα λοιπόν με το τι συμβαίνει στην ε, Ισπανία με τις φράουλες, εδώ στην Βόρεια ε, Ελλανδία ε, προτιμώνται γυναίκες με παιδιά για να μπορούν να εργάζονται πολύ περισσότερο. Οι γυναίκες αυτές δεν ξέρουν καλά αγγλικά, έχουν, έχουν συναδέλφισες μέσης ηλικίας, και έτσι αναγκάζονται να δουλεύουν μέχρι πολύ αργά το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα. Ε, προσλαμβάνονται υπό διάφορε περιστάσει και συνθήκε ε, ανάλογα με το σε ποια φάση τη ζωή του βρίσκονται. Και αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε ότι οι γυναίκε εδώ προσπαθούν να ενσωματωθούν στην κοινωνία, να μάθουν αγγλικά. Κάποιες πηγαίνουν και στην εκκλησία, ε, μελετούν, ε, μαθαίνουν αγγλικά, αλλά ε, πολλές φορές τους απαγορεύεται αυτό. Γιατί αν πάει στην, στην, στην, στο σχολείο στις 7 το πρωί, η βάρδια της θα πάει μέχρι πάρα πολύ αργά. Και τους λένε οι εργοδότες, όχι εδώ έχεις έρθει για να δουλεύεις, όχι για να πας να μάθεις αγγλικά. Άρα δεν διευκολύνονται οι γυναίκες αυτές ούτε προς την ένταξή τους. Αντίθετα, ε, με αυτόν τον τρόπο και με αυτές τις συνθήκες στις οποίες αναγκάζονται να ζουν, ε, διαιωνίζεται αυτή η κοινωνική του περιφερειοποίηση. Βλέπουμε επίσης ότι οι υποδομέ που υπάρχουν δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μεταναστριών αυτών. Ε, υπάρχει, δεν υπάρχουν πολλές φορές, για παράδειγμα, ούτε τουαλέτες. Σε ένα εργοστάσιο μάλιστα υπήρχε, υπήρχαν δύο διαλύματα που προβλέπονταν, 20 λεπτά υποτίθεται, 11, 11 λεπτά ήταν ε, στην πραγματικότητα και πάντοτε υπήρχε μόνο μία τουαλέτα και υπήρχαν τεράστιες σουρές. Οι γυναίκες δεν μπορούσαν να πάνε στην τουαλέτα δηλαδή, στο διάλειμμα τους. Πάρα πολύ σκληρή δουλειά λοιπόν, ήλιο με ήλιο, ε, κουβαλάς μήλα ε, εκατοντάδες κυβότια τελάρια, τελάρα ε, μέχρι που πονάει το σώμα σου πολλές φορές ε, μέχρι τις 6-8 το βράδυ ή και ακόμα και τις 11 το βράδυ και μετά 6 ώρα το πρωί ξεκινάει ξανά η καινούρια βάρδια. Είναι σκλαβιά κανονική. Δεν έχω ξαναζήσει λέει, μια γυναίκα ποτέ τέτοια συνθήκη. Στην αρχή έλεγα εντάξει, αφού μπορούν και άλλε γυναίκε να το κάνουν, θα το κάνω κι εγώ, θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Ε, βλέπουμε δηλαδή μια παρέτηση των ανθρώπων, μια αποδοχή μυρολατρική των συνθήκων εντός των οποίων έχουν ε, βρεθεί αυτές οι γυναίκες. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρά θέματα. Μία από τις δυσκολίες λοιπόν είναι ότι η αγροτική εργασία είναι ένας τομέας στον οποίο μπορεί να υπάρχει μεγάλη συμπίεση των μισθών και μεγιστοποίηση των ε, κερδών είναι πιο ακριβό να αγοράσει κανείς ένα μηχάνημα από το να εκμεταλλευτεί ε, μια ε, υποαμοιβόμενη γυναίκα. Και παρά το γεγονός λοιπόν ότι ε, και είναι χαρακτηριστικό ότι παρότι είναι τόσο χαμηλή η μισθή είναι πάλι υψηλότερη από ό,τι στις χώρες καταγωγής τους. Το ηθικό και νομικό ερώτημα λοιπόν είναι γιατί οι γυναίκες αυτές μετανάστριες καταλήγουν να ζουν σε συνθήκες που είναι συγκρίσιμες με, με τους ε, μετανάστες χωρίς χαρτιά στις ΙΠΑ, για παράδειγμα. Πώς το σύστημα μας έχει επιτρέψει να φτάσουμε σε, αυτή την κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν ε, η νομοθεσία να εφαρμοστεί ε, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η αυτονομία που έχουν οι γεωργοί προστατεύεται πάρα πολύ. Άρα το ερώτημα είναι πώς ακριβώς θα ξεπεράσουμε αυτό το, αυτό το τεράστιο σύνολο προβλημάτων που υπάρχουν. Σημαντική προσοχή πρέπει να δοθεί λοιπόν στη μεταποίηση τροφίμων ε, αλλά και σε όλους τους άλλους αγροτικούς ε, και γεωργικούς κλάδους όπου διαπιστώνεται τεράστια εκμετάλλευση γυναικών. Εγώ σας ευχαριστώ. Thank Και τώρα συζήτηση τα μέλη ε, της Επιτροπής η Ράτσε Γαρθία Πέρεθ. Καλημέρα σας. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλες τις ε, προσκεκλημένες που συμμετέχουν στην ακρόαση αυτή για την κατάσταση των ε, μεταναστευτριών στις αγροτικές περιοχές. Ακούσαμε τρεις παρεμβάσεις στην αρχή και φαντάζομαι και στη συνέχεια θα ακούσουμε τα ίδια. Είναι πολύ γνωστή αυτή η πραγματικότητα σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια με τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας λόγω της γεωργικής δραστηριότητας σε κάθε χώρα. Η πραγματικότητα όμως είναι ίδια. Υπάρχει ένας ευάλωτος τομέας, η γεωργία, όπου είναι πολλοί εργαζόμενοι και πολλές φορές μετανάστες και πάντα όταν αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ευάλωτους τομείς στο εσωτερικό του κάθε κλάδου υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία λόγω του φύλου. Δηλαδή μπορεί να είναι ο κλάδος ιδιαίτερος με δυσκολίες και οι μετανάστες να έχουν πάντα δυσκολίες. Όταν είσαι όμως μετανάστρια έχεις πολύ περισσότερα προβλήματα. Ακούσαμε ποια είναι αυτά. Πέρυσι είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ τη Ραγκούσα. Πήγα και είδα και την Φρανσέσκα και επισκεφθήκαμε τις γυναίκες αυτές και μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα και έρχονται σε επαφή και παρέχουν και βοήθεια στις εργαζόμενες μετανάστριες, αλλά συναντήσαμε και γεωργικές ε, οργανώσεις. Επισκεφτήκαμε εκμεταλλεύσεις δηλαδή και χώρος ε, που είχαν ειδικά προγράμματα φροντίδας στις γυναίκες και είναι σημαντικό να το λέμε και αυτό ότι υπάρχουν και τέτοια και υπάρχουν και γεωργικές επιχειρήσεις ε, που ασχολούνται με την παροχή στήριξης και βοήθειας στις γυναίκες αυτές και το ρυθμίζουν σωστά. Εν πάση περιπτώσει, γενικά ισχύει αυτό που είπατε. Εκμετάλλευση τις ευάλωτες θέσεις των γυναικών, δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες, όπως μπορεί να είναι η εκπαίδευση, το σχολείο των παιδιών, ακόμα, ακόμα και για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση και ανατριχιάζουμε ακούγοντας τι αναγκάζονται να ζουν αυτές οι γυναίκες. Θέλω λοιπόν να ξέρω το έργο των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με τις γυναίκες αυτές, αλλά και να σας αναφέρω και κάτι, μια καταγγελία. Οι πολιτικές λιτότητας και οι περικοπές ε, είχαν μεγάλες επιπτώσεις γενικά στη ζωή αλλά και στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί εκεί στη Ραγκούσα όταν συναντηθήκαμε με τις αρχές τοπική αυτοδίκησης, μας είπαν ότι είναι πάρα πολύ πενιχρά τα μέσα που έχουν οι ανθρώπινοι πόροι στην επιθεώρηση εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλό είναι να έχουμε νόμους ε, που να προστατεύουν αυτές τις εργαζόμενες, αλλά χρειάζονται και έλεγχοι. Επιθεώρηση εργασίας ισχυρή για να μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες. Και αν έχεις έναν επιθεωρητή εργασίας σε μια γεωγραφική περιοχή με 500 ας πούμε περίπου γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τι να κάνει ο άνθρωπος ο ένας και πώς να ελέγξει και πώς να επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες. Κάτι που μου τράβηξε την προσοχή είναι αυτό που μας είπαν ορισμένοι εκτιματίες. Ε, δεν έπεσαν από τα σύννεφα. Μα είπαν ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο και το γνώριζαν. Δεν ήταν κάτι αποσπασματικό. Και υπάρχουν και επιχειρηματίε που αναγνωρίζουν αυτήν την πραγματικότητα, το ξέρουν ότι συμβαίνει. Και υπάρχουν και κάποιοι που το αντιμετωπίζουν και κάνουν πολύ καλή δουλειά και σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων λοιπά Και μας είπαν ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε οι πρώτοι ενδιαφερομένοι να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί δημιουργείται μια δημόσια εικόνα και δημιουργούνται τέτοιες εντυπώσεις που είναι εις βάρος ε, και της ε, δουλειάς εδώ και των προϊόντων και της παραγωγής μας. Τελειώνω. Επιθεώρηση. Ε, χρειαζόμαστε ελεγκτές μπορεί να έχουμε νομοθεσία που προστατεύει τις γυναίκες αυτές, αλλά θα πρέπει να επιβάλλει την νομοθεσία. Και οι επιθεωρητές να έχουν στη διάθεσή τους ό,τι χρειάζονται για να μπορούν να το κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Επίσης, θα πρέπει να στηρίξουμε τις οργανώσεις που συμπαραστέκονται στις γυναίκες αυτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να τονίσουμε και να διατρανώσουμε την ανάγκη στήριξης αυτών των οργανώσεων, που πραγματικά κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και υποκαθιστούν αυτό που θα έπρεπε να κάνει η κρατική μηχανή, που δεν το κάνει. Συντονισμός χρειάζεται, στήριξη των οργανώσεων, στήριξη των επιθεωρήσεων εργασίας και το γεγονός και μόνο ότι γίνεται σήμερα εδώ αυτή η ακρόαση ε, αποτελεί απόδειξη ε, ότι υπάρχει ευαισθησία και ανταπόκριση για να βελτιωθεί η κατάσταση. Και εδώ μιλώ για όλη τη γεωργία για τους μετανάστες εργαζομένους στην ε, Γεωργία και ιδιαίτερα τις γυναίκες, τις μετανάστριες που είναι όλο και πιο ευάλωτες και ακόμα περισσότερο. Τελειώνω λοιπόν. Σας ευχαριστώ που ήρθατε να μας ενημερώσετε για αυτή την κατάσταση και η σοσιαλιστική ομάδα πραγματικά θα συνεχίσει και δεσμέγεται γι' αυτό να εργάζεται προς την κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας της ζωής αυτών των εργαζομένων γυναικών. Ευχαριστώ κύριε Αγκαρθία Πέρες. Tack. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω σουηδικά. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τις προσκεκλημένες μας, οι οποίες πραγματικά μας κάνουν κάποιες πολύ καλές παρουσιάσεις. Γνωρίζουμε ότι όλα αυτά λαμβάνουν χώρα. Όταν βλέπει κανεί φωτογραφίε, πραγματικά η κατάσταση αλλάζει. Εγώ από το 2009 ασχολούμαι με την εμπορία ανθρώπων και το 2011 ασχολήθηκα με την κατάρτιση της κοινοτική νομοθεσίας κατά της εμπορίας ανθρώπων. Μια νομοθεσία που βέβαια από μόνη τη δεν μπορεί να επιλύσει όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με την νομοθεσία αυτή, να την επικαιροποιήσουμε, να την αναθεωρήσουμε για να καλύψουμε και όλες αυτές τις νέες εκφάνσεις του προβλήματος που βλέπουμε τώρα. Δεν θυμάμαι ακριβώ το όνομά σα. Μα κάνετε εσεί πάντω την πρώτη παρουσίαση με τι φωτογραφίε και μα δείξατε τη φωτογραφία από το μικρό αυτό κοριτσάκι που είχε ακολουθήσει τη μητέρα του. Όλε αυτέ οι γυναίκε οικειοθελώ έρχονται αποφασίζουν συνειδητά να έρθουν να εργαστούν, αναγκάζονται τροποντινά γιατί δεν έχουν ε, καθόλου χρήματα στη χώρα τους, στη Ρουμανία. Όταν φτάνουν όμως στις περιοχές αυτές της Ιταλίας που μας δείξατε, αυτόματα αποτελούν θύματα εμπορίας ανθρώπων. Είναι πραγματικά θύματα και ως τέτοια θα πρέπει να αναγνωριστούν. Γιατί όχι μόνο εργάζονται για πενταροδεκάρες πραγματικά, αλλά γιατί πραγματικά πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Μας είπατε ότι ε, αναγκάζονται να αφήσουν ανοιχτή την πόρτα το βράδυ όταν κοιμούνται για να μπορεί να μπαινοβγαίνει ελεύθερα ο εργοδότης. Ε, καταλαβαίνετε επίση ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε όχι μόνο τι γυναίκε τι ίδιε, αλλά και τα παιδιά του, γιατί και τα ίδια πέφτουν θύματα σεξουαλική κακοποίηση. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε μια τέτοια κατάσταση στην Ευρώπη σήμερα. Όλα τα κράτη-μέρη φέρουν τεράστια ευθύνη και οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες τους περγάζονται στο εξωτερικό δεν θα αποτελούν θύματα κακοποίησης εκμετάλλευσης. Είναι τεράστια ευθύνη που μας βαρύνει όλους. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω το ακόλουθο ερώτημα. Είπατε πριν από λίγο ότι οι γυναίκες αυτές πληρώνονται 10 με 20 ευρώ την εβδομάδα. Θεωρείτε ότι πληρώνονται λιγότερο από τους άντρες, ακόμα και όταν κάνουν την ίδια δουλειά με αυτούς. Και πόσες γυναίκες ε, πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης κατά αυτόν τον τρόπο. Θα θέλαμε να έχουμε λίγο περισσότερα αριθμητικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Νόχελ και μετά οι υπόλοιποι. Θέλω να αναφερθώ σε κάτι που είπε η προλαλή και μας απασχολεί ε, και στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ότι έρχονται εθελοντικά, είπατε. Εθελοντική είναι και η πορνεία καμιά φορά τα και τα συζητάμε. Εθελοντική είναι και η παρένθετη μητέρα. Εθελοντική είναι και η δωρεάν οργάνων. Και εθελοντική είναι και η εργασία σε τέτοιες θέσεις εργασίας που κανένας δεν τις θεωρεί επιθυμητέ. Γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση λοιπόν σε βάθο για το εθελοντικό όλων αυτών των υποθέσεων. Και καμιά φορά και στα ίδια μας τα κόμματα και στη δική μας ε, παράταξη ε, είμαστε κατακαιρματισμένοι. Υπάρχει το δικαίωμα της γυναίκα να αποφασίσει τι θα κάνει με τη ζωή της, αλλά σε κανένα από αυτά που σας ανέφερα δεν βλέπω ε, κανένα εθελοντικό στοιχείο. Όλα αυτά δεν είναι καθόλου εθελοντικά. Όλα αυτά είναι αποφάσεις που αναγκάζονται να παίρνουν οι γυναίκες γιατί είναι στριμωγμένες στον τοίχο και υφίσταται μία πίεση για να βγουν από μία κατάσταση και είναι το μη χειροβέλτιστο. Δεν μπορεί, ε, μπορεί να είναι μπρο γκρεμό και πίσω ρεύμα το, το, το, το εθελοντικό. Υποστηρίζω λοιπόν τις προαλήσεις ε, και την κυρία Χέτ που μίλησε μέσα πριν από μένα δούμε. Πολύ ωραίο αυτό που είπατε για τη Ρουμανία, για την ενημέρωση, για τη μαζική ενημέρωση των γυναικών και ποντάρετε εκεί. Είναι πολύ σημαντικό τουλάχιστον να ε, γνωρίζουν είναι αρκετά δυσάρεστο ότι τους βγάζει ανάγκη ε, σε αυτή την κατάσταση, αλλά τουλάχιστον να γνωρίζουν τι τις περιμένει. Και άνδρες και γυναίκες, γιατί δεν φταίνε μόνο οι άνδρες, οι ένοχοι να πηγαίνουν και φυλακοί όταν εκμεταλλεύονται την ανάγκη και την φτώχεια ε, και να πλουτίζουν. Δεν αρκεί να τους ε, επιβάλλουμε πρόστιμα και κυρώσεις ε, ή να τους φοβερίζουμε. Εδώ πατάσουμε το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών και τη διακίνηση εκμετάλλευση των ανθρώπων δεν θα πρέπει ε, να το πατάσουμε. Εγώ γενικά είμαι ήπια στους τόνους, αλλά ε, εδώ χρειαζόμαστε πάρα πολύ σαφείς νόμους. Όποιος εκμεταλλεύεται την απόγνωση και την ανάγκη του άλλου είναι δουλέμπορος όσο και αν υποτίθεται ότι τον αμείβει τον άλλον. Και θα πρέπει να πείπτει και ράβδος, όχι μόνο πρόστιμα και φυλακή. Θα πρέπει η Ευρώπη να είναι φάρος. Να... Χρειαζόμαστε νομοθεσία. Δεν λέω, δεν μπορούμε να την επιβάλλουμε παντού, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένας γνώμονας. Τι είναι σωστό και τι είναι λάθος να το ξεκαθαρίζει ο νόμος. Είτε πρόκειται για πρόσφυγες που είναι εδώ και δεν έχουν κανένα καθεστώς, είτε πρόκειται για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μένα δεν υπάρχει καμία διαφορά. Για μένα αυτό είναι πραγματικό δούλεμπόριο και πατάσετε μόνο με πάρα πολύ ε, βαρύες κυρώσεις. Ευχαριστώ κύριε Νόχη. Η κυρία Ζάνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ακρόαση αυτή. Ήταν πραγματικά είναι πολύ ευαίσθητο και πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Πρόκειται για μια πραγματικότητα από την οποία δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Είναι μια κοινωνική πραγματικότητα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να συζητήσουμε την πραγματικότητα αυτή με του πολίτε μα το συντομότερο δυνατό και όχι απλώ να ευαισθητοποιήσουμε κάποιε αρχέ. Αντίθετα, να ασκήσουμε πίεση στις αρχέ σε τοπικό επίπεδο, σε αυτέ τι αγροτικέ περιοχέ όπου ε, εμφανίζονται αυτές οι καταστάσεις όπου υπάρχουν γυναίκες που δουλεύουν σε αγροτικές δουλειές και γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Φυσικά ε, στη Ρουμανία και σε ολόκληρο τον κλάδο της γεωργίας, σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που ε, γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευση, που υφίστανται εκμετάλλευση και είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε αυτές τις, τις γυναίκες. Ως Ρουμάνα Ευρωβουλευτής όμως έχω καθήκον και υποχρέωση να προστατεύσω ε, και τα δικαιώματα των γυναικών ε, εργατριών ε, που εργάζονται ε, στη γεωργία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω στη δική μας περίπτωση στην Ιταλία και στην Ισπανία. Γι' αυτό και είναι απόλυτα αναγκαίο άμεσα όλα τα κράτη-μέλη να αναλάβουν άμεσα δράση και να σταματήσουν να ανέχονται αυτή την κατάσταση. Πρέπει να, κατα... να καταγγείλουμε βεβαίως και να διώξουμε όλες τις καταστάσεις βίας που υφίστανται αυτές οι γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές, ιδίως στην Ιταλία και στην Ισπανία, δεν εργάζονται σε αξιοπρεπείς συνθήκες, δεν έχουν εξοπλιστεί συνθήκε εργασία και διαβίωση, δεν έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία ε, ούτε καν να μεταφέρονται από τον τόπο στον οποίο διαμένουν μέχρι τα θερμοκήπια στα οποία εργάζονται. Τα παιδιά του δεν μπορούν να πάνε σχολείο για τον ίδιο λόγο, γιατί δεν υπάρχουν ε, μεταφορικά μέσα μεταξύ των χώρων εργασία του και των χώρων διαβίωσή του. Γιατί δεν προβλέπεται και δεν παρέχονται μεταφορικά μέσα στι γυναίκε αυτέ. Δεν υπάρχουν σχολεία ε, και μάλιστα διαπιστώνονται γίνονται και πάρα πολλές περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Όλα αυτά πρέπει να αναγνωριστούν ως αυτό που είναι, μια κοινωνική ε, παρενόχληση ε, σοβαρότατης μορφής. Δεν γίνεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πρέπει από τα λόγια να περάσουμε στις πράξεις τώρα. Βεβαίως, η μισή τους είναι το, το πρώτο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι γυναίκες αυτές έρχονται σε αυτέ τι αγροτικέ περιοχέ όχι γιατί δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν, αλλά γιατί χρειάζονται λεφτά. Βεβαίω, όταν δεν εξασφαλίζεται η έγκαιρη αμοιβή του, αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στι οικογένειε τι οποίε υποτίθεται ότι έχουν πάει να υποστηρίξουν, έχουν πάει στι αγροτικέ περιοχέ αυτέ για να υποστηρίξουν στι χώρε καταγωγή του. Και αυτό είναι ο λόγο που οι γυναίκε αυτέ επιτρέπουν στου άλλου να του συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, να τι μεταχειρίζονται με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι σε οικονομική ανάγκη οι γυναίκε αυτέ. Άρα έχουμε ένα, ένα, ένα, ένα πολυπλόκαμο σύστημα το οποίο τι καταπιέζει αυτέ τι γυναίκε. Είναι οικονομική ανάγκη, κοινωνικό αποκλεισμό, έλλειψη μεταφορών και αυτό είναι ένα, ένα θέμα το οποίο βεβαίω πρέπει να αντιμετωπιστεί και νομοθετικό για να προστατεύονται οι γυναίκε αυτέ και να βεβαίω να εξασφαλίζεται και η, η εφαρμογή τη νομοθεσία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην εμπειρογνώμονα από το θεματικό τμήμα ε, για τα δικαιώματα των πολιτών και τις συνταγματικέ υποθέσεις. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Σούρμπα και μετά στην κυρία Παλόμπο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ πέρα και μπορούμε να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη μας. Εγώ θα σας παρουσιάσω το πρώτο τμήμα και η συνάδελφος η κυρία Παλούμπο το δεύτερο τμήμα. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, δεν μπορούμε να καλύψουμε όλα τα ζητήματα τα οποία θίγουμε με την έκθεσή μας, αλλά προσβλέπουμε και σε μια θετική συζήτηση μαζί σας. Να παρουσιάσω καταρχάς τους βασικούς στόχους της μελέτης αυτής. Θέλουμε μέσω μιας ποιοτική προσέγγισης να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν την απασχόληση των ε, μεταναστριών γυναικών στις γεωρικές εκμεταλλεύσεις και ασχοληθήκαμε κυρίως με την περίπτωση της Ιταλίας και της Ισπανίας. Θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι διαρθρωτικές συνθήκες και συγκεκριμένες καταστάσεις που βιώνουν οι γυναίκες στις περιοχές αυτές και να δούμε εν συνεχεία πώς μπορούν να ληφθούν υπόψη πολιτικές που θα μπορούσαν να στραφούν κατά της ε, εργασιακής εκμετάλλευσης αλλά και των φαινομένων δουλείας ή ακόμα και των φαινομένων εμπορίας ανθρώπων. Κάνουμε συνεχεία κάποιες συστάσεις για τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διάσταση της ισότητας των φύλων. Ξεκινήσαμε από ένα συγκεκριμένο νεολογικό πλαίσιο, στο κέντρο του οποίου θέσαμε τον ευάλωτο χαρακτήρα της κατάστασης των γυναικών βάλτος αυτός χαρακτήρας δεν έχει να κάνει μόνο με τα γενή χαρακτηριστικά των γυναικών και της κατάστασής τους, αλλά ένας ευάλωτος χαρακτήρας που έχει να κάνει με τον πιο τρωτό προφίλ που έχουν οι γυναίκες εξαιτία των καταστάσεων που ζουν. Θέλαμε ουσιαστικά να δούμε πιο συγκεκριμένα την κατάσταση των γυναικών και των παιδιών και αυτό που μας απασχολεί όλος ιδιαιτέρως είναι ο ευάλωτος χαρακτήρας που προκύπτει από συγκεκριμένε καταστάσεις που επιβάλλονται στις γυναίκες λόγω εξωτερικών δομικών παραγόντων. Λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν την ε, κατάσταση των εργαζόμενων μεταναστρατιών στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες ε, πολλές φορές αντιμετωπίζουν μια διατομιακή διακριτική μεταχείριση και που αποκλείονται όχι μόνο επειδή είναι γυναίκες, αλλά λόγω του καθεστώτος του μετανάστη που έχουν, το γεγονός ότι βρίσκονται εκτό τη κοινωνία, εκτός του συστήματος κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό επιτείνει ακόμα περισσότερο την ευάλωτο χαρακτήρα των γυναικών αυτών όπως ορίζεται στην Οδηγία 36 του 2011. Εκεί πέρα ο ευάλωτο χαρακτήρας ορίζεται ως η κατάσταση των γυναικών εκείνων, των ανθρώπων εκείνων που δεν έχουν εναλλακτικέ πέρα από το να αποδεχθούν τελικά την κατάσταση την οποία βιώνουν. Πολλές φορές οι γυναίκες αυτές αναγκάζονται να αποδεκτούν συγκεκριμένε καταστάσεις, ακόμα και αν αυτές εμπεριέχουν τελικά κακοποίηση ή εκμετάλλευση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η οδηγία αυτή αναφέρεται και στην έννοια της σύμφωνης γνώμης, της οικιοθελούς αποδοχής των γυναικών αυτών. Μας ενδιαφέρει να δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών ροών καθώς επίσης και των συνθήκων εργασίας της γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Όσον αφορά τη μετανάστευση καταρχάς, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν πάντα ασφαλείς και νόμιμοι οδοί για να φτάνει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουμε παράτυπες μορφές μετανάστευσης εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε πολλές φορές ότι οι μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίθενται κατά τον ίδιο τρόπο σε εκμετάλλευση και κακοποίηση με τους μετανάστες που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι υπάρχουν θέσεις απασχόλησης που καλύπτονται από γυναίκες στον γεωργικό τομέα εκεί ακριβώς που δεν ρυθμίζονται ακριβώς συνθήκες εργασίας και οι γυναίκες κατά αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουν συγκεκριμένε ε, μορφές ε, τροτότητας που έχουν να κάνουν περισσότερο με τον ε, ευάλωτο χαρακτήρα που έχει να κάνει με το γυναικείο φύλλο. Επίσης, πολλές φορές βλέπουμε ότι το δικό τους το νομικό καθεστώς, καθεστώς το γεγονός ότι ζουν μόνες τους, τις καθιστά ακόμα πιο ευάλωτες στα πλαίσια του γεωργικού τομέα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει όλο και περισσότερο ένα συγκεκριμένο μοντέλο παραγωγής το οποίο το βλέπουμε όλο και περισσότερο στο γεωργικό τομέα το οποίο ουσιαστικά στρέφεται όλο και περισσότερο στην απασχόληση γυναικών, στην εκμετάλλευση των γυναικών ή ακόμα και στην κακοποίηση των γυναικών. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να περάσουμε πλέον πέρα από τις βασικές προτεραιότητες που έχουμε στην κοινή γεωργική πολιτική που είναι ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα σε μια πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη της και τις εργασιακές συνθήκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα εξακολουθήσουμε να βλέπουμε ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά θα υποτάσει όλο και περισσότερο τις γυναίκες και ουσιαστικά θα τις χρησιμοποιεί ως φτηνά εργατικά χέρια. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει εδώ πέρα να ασχοληθούμε όλο και περισσότερο με το ζήτημα των ε, μεταναστών που εργάζονται στο γεωργικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε ακριβώς πώς οι σχέσεις ισχύως, οι σχέσεις εξουσίας επηρεάζουν κυρίως την κατάσταση των γυναικών. Βλέπουμε επίσης ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αναλυτικά δεδομένα μεμονωμένα για τη θέση των γυναικών στο γεωργικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις τώρα μελέτες που κάναμε στην Ισπανία και την Ιταλία. Επιλέξαμε τις δύο αυτές χώρες γιατί έχουν γίνει όλο και περισσότερο σημαντικοί προορισμοί για μετανάστες που έρχονται όχι μόνο πλέον από τη Βόρεια Αφρική αλλά και από τις ανατολικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ιδίως στην Ιταλία και στην Ισπανία ασχοληθήκαμε με τις περιπτώσεις εκείνες των ε, μεταναστριών γυναικών οι οποίες απασχολούνται στο γεωργικό τομέα, όπου ο αριθμός τους πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όσον αφορά την Ιταλία, ασχοληθήκαμε με την επαρχία της Ραγκούσα, κυρίως για τους λόγους που παρουσίασε η Φραντσέσκα. Στην ε, Ραγκούσα αρχίσαμε να εργαζόμαστε το 2013. Επίσης ασχοληθήκαμε και με άλλες περιοχές Ιταλίας όπου έχουμε εργαζόμενες από την Αφρική και άλλες περιοχές όπου οι γυναίκες ζουν πραγματικά σε γκέτο ή υφίστανται σεξουαλική εκμετάλλευση. Όσον αφορά την Ισπανία ασχοληθήκαμε με την επαρχία της Σουέλβα και αυτή αναφέρθηκε πριν από λίγο. Είδαμε την παραγωγή φραουλών και με την περιοχή της Αλμέιρα που θεωρείται πραγματικά τον αποκαλούν πολλές φορές το πλαστικό πέλαγος, μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν εκεί πέρα τόσες γεωρικές εκμεταλλεύσεις και πάρα πολλά θερμοκήπια, στα οποία απασχολούνται πάρα πολλές γυναίκες. Όσον αφορά την ε, Ιταλία, βασιστήκαμε στην δική μας τη μελέτη, όσον αφορά την Ισπανία βασιστήκαμε και σε κάποιες πρώτερες μελέτες που είχαν γίνει. Στα πλαίσια των ε, ερευνών αυτών θελήσαμε να δούμε καταρχάς ποιες είναι οι πολιτικές οι οποίες χρησιμοποιούνται όσον αφορά την ε, εποχική μετανάστευση, την κυκλική μετανάστευση και επασχόληση των γυναικών στο γεωργικό τομέα. Συστήματα δηλαδή τα οποία έχουν προκύψει και αποκαθιστούν τις γυναίκες όλο και πιο ευάλωτες. Στην Ισπανία υπάρχουν δύο διαφοροποιημένα επίπεδα. Έχουμε εποχικές μετανάστρες κυρίως από το Μαρόκο, γιατί προφανώς η εκμετάλλευση και η κακοποίηση έχει να κάνει μόνο με την Ανατολική Ευρωπαϊκή Ένωση και ασχοληθήκαμε βέβαια και με τις μετανάστριες, τις εργαζόμενες στον τομέα του γεωργικού, στον γεωργικό κλάδο που προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη. Στην περιοχή της Σουέλβα έχουμε γυναίκες από τρίτες χώρες ή και από την Ανατολική Ευρώπη που έχουν συμβάλει πάρα πολύ στο να αντικατασταθεί το γεωργικό δυναμικό το οποίο υπήρχε στην περιοχή εκείνη, προκειμένου να έχουμε πλέον εργαζόμενους οι οποίοι θα αποδέχονται όλο και μεγαλύτερη ευελιξία. Κατά αυτόν τον τρόπο είχαμε έναν κατακαιρματισμό της αγοράς εργασίας στο γεωργικό τομέα με βάση το φύλλο, με βάση την εθνοτική καταγωγή και το, καθεξής και βλέπουμε πολλές φορές ότι χρησιμοποιούνται μέσα τα οποία καθιστούν την εργασία όλο και πιο ευέλικτη και όλο και πιο κατακαιρματισμένη. Στα πλαίσια των ερευνών αυτών είδαμε ότι στην Ιταλία και στην Ισπανία οι μετανάστρες εργαζόμενες εντός και εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν επαχθείς εργασιακές συνθήκες, αυτές που ακούσαμε σήμερα, πολύ συχνά είναι ανειδίκευτες και πιο νέες από ό,τι έχουμε σε άλλους τομείς και έχουν λιγότερους προσωπικούς πόρους για να καταφέρουν τελικά να αντιταχθούν στις συνθήκες εκμετάλλευσης οι οποίες αποδέχονται, ζουν απομονωμένες και αυτό το καλύψαμε και στην Αλμέιρα, στην Ραγκούσα ή και σε άλλες περιοχές έχουμε πραγματικά μια γετοποίηση των γυναικών αυτών. Αυτό το είδαμε και στην Ουέλβα. Εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την εργασία τους και από τους εργοδότες τους. Και το γεγονός ότι έχουν και εξαρτώμενα μέλη τις καθιστά ακόμα πιο ευάλωτες. Το είδαμε αυτό και στην περίπτωση της Ραγκούσα το κάλυψε αυτό η Φραντσέσκα στην παρουσίαση που έκανε. Τώρα όσον αφορά τις γυναίκες από τη Ρουμανία που εργάζονται στην Ραγκούσα, είδαμε ότι οι γυναίκες αυτές υφίστανται πάρα πολύ συχνά εκβιασμούς, εξαναγκασμούς, σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση και κατά αυτόν τον τρόπο τους ασκείται μια πολύ έντονη ψυχολογική πίεση. Και αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ότι ε, ακριβώς επειδή τελούν σε καθεστώς ψυχολογικής πίεσης και εξάρτησης, οι γυναίκες αυτές τελικά δεν καταφέρνουν να καταγγείλουν τα κακό και δεν ε, μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο να κινηθεί μια ποινική δίωξη κατά των ε, παραβατών. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα γενές πλέον σύστημα το οποίο έχει ριζώσει στις περιοχές αυτές και το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε νέες μορφές καταναγκαστικής εργασίας ή ακόμα και δουλείας και σε άλλες έρευνες βλέπουμε ότι αντίστοιχα φαινόμενα έχουμε και στην Ουέλβα της Ισπανίας, αλλά και στις δύο χώρες πάντως έχουμε περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών, οι οποίες μπορεί να μην εμπλέκονται άμεσα στο γεωργικό τομέα, και οι οποίες απλώς ζουν σε γκέτο ή σε απομονωμένες γεωργικές περιοχές. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, είδαμε ότι οι γυναίκες οι οποίες ζουν σε αυτά τα γκέτο, χωρίς να έχουν καμία πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες στέγασης, βρίσκονται πάλι σε μια πάρα πολύ ευάλωτη θέση και πάρα πολύ συχνά υφίστανται σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση. Μέσω της δικής μας της μελέτης και μέσω των άλλων μελετών βλέπουμε ότι καταρχάς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους διαρθρωτικούς εκείνους παράγοντες που καθιστούν τις γυναίκες πιο ευάλωτες. Πρέπει δηλαδή να αναλύσουμε περισσότερο τις συνθήκες εργασίας στον γεωργικό τομέα. Ολοκληρώνοντας το σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Λετίτσια η οποία θα αναφερθεί στο τμήμα εκείνο της έκθεσης που αναλύει περισσότερο το εφιστάμενο νομικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Good afternoon. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω τώρα το δεύτερο τμήμα της μελέτης μας και συγκεκριμένα στην μελέτη μας αφιερώσαμε ε, ένα τμήμα αυτής στην ανάλυση του διεθνούς και του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της καταναγκαστικής εργασίας. Ιδίως ως προς το διεθνές δίκαιο ε, ε, εξετάσαμε τους ορισμούς ε, για την καταναγκαστική εργασία που έχει που ενσωματωθεί στην, συγκεκριμένη, στην σχετική συνθήκη και βλέπουμε ότι ο, ο, δεν υπάρχει ακόμη επαρκής σαφήνεια, διάκριση μεταξύ αυτών των του, των, ενιών του τράφικινγκ και της καταναγκιστικής εργασίας και αυτό προέκυψε και σε πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ιδίως όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και το τράφικινγκ ε, έχουμε την συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005 για την καταπολέμηση του τράφικινγκ ε, το οποίο έχει ε, ε, μια προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ταυτόχρονα ε, αναδεικνύεται ότι η σύμβαση αυτή ε, είναι σημαντικό μέσο και μηχανισμός για την μη ποινικοποίηση των θυμάτων του τράφικινγκ. Αυτές οι αρχές και της, και της απροϋπόθετης ε, βοήθειας και αυτό επιβεβαιώθηκε και στο σχετικό πρωτόκολλο του Διεθνούς ε, ε, Οργανισμού Εργασίας σχετικά με την καταναγκαστική εργασία και αναδεικνύουμε πως το πρωτόκολλο 29 ε, επίσης υιοθετεί μια τέτοια προσέγγιση βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά την καταναγκαστική εργασία. Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά μέσα νομοθετήματα, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στην ε, οδηγία 2011 36 αναδεικνύονταν πως αυτή η οδηγία αποτέλεσε ένα σημείο καμπής ε, όσον αφορά την ευρωπαϊκή στάση απέναντι στο ζήτημα, λαμβάνοντας υπόψη μια προσέγγιση που ενισχύει περισσότερο τη διάσταση του φύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, βασική αρχή της απροϋπόθετης αρρωγής και της μη ποινικοποίησης, μη δίωξης των θυμάτων, ε, ε, διαπιστώσαμε ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί αυτή, οι, αυτές, δεν έχουν ενσωματωθεί επαρκώς ακόμα αυτές οι δύο αρχές στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Φαίνεται ότι η οδηγία αυτή, η 2011-36, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί επαρκώς σε πολλά κράτη-μέλη, ιδίως όσον αφορά την προστασία και την αρρωγή που παρέχεται στα θύματα. Όσον αφορά άλλα νομοθετικά ευρωπαϊκά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, καταπολέμηση της ε, ε, εκμετάλλευσης και το τράφικινγκ. Δεν έχω χρόνο να σας τα πω όλα, αλλά θέλω να επισημάνω κάποια στοιχεία που σχετίζονται με την Οδηγία 2014-36 για τους εποχιακούς εργαζόμενους και στη μελέτη μας αναδεικνύουμε πώς η οδηγία αυτή περιλαμβάνει τη δυνατότητα των εργαζομένων να αλλάξουν ε, εργοδότη. Ωστόσο αυτή η διάταξη δεν είναι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη και όπως προκύπτει από, την, ε, από τις μελέτες μας, ιδίως στην ε, Ισπανία, μόνο μερικώς περιορίζει η διάταξη αυτή τον ευάλωτο χαρακτήρα των εργαζομένων γυναικών. Τέλος, θέλω επίσης να αναφέρω ότι εξετάσαμε την ενωσιακή νομοθεσία για την απόσπαση των εργαζομένων και διαπιστώσαμε ότι δεν ε, αντιμετωπίζει επαρκώς ε, ε, τη, τα φαινόμενα κοινωνικού dumping και γι' αυτό και η Κομισιόν πρόσφατα πρότεινε αναθεώρηση της οδηγίας 96-78 για να θεσπιστούν καλύτεροι κανόνες για την ανταγωνιστικότητα και καλύτερη εξισορρόπησή τους με τα κοινωνικά δικαιώματα. Πέρα λοιπόν από τα ευρωπαϊκά νομοθετήματα για την καταπολέμηση του τράφικινγκ και της εκμετάλλευσης, εξετάσαμε λοιπόν το, τη συνολική εικόνα ε, λαμβάνοντας υπόψη και τις πολιτικές για τη μετανάστευση. Και εδώ αναδεικνύουμε ότι η καινοτόμα ε, ε προσέγγιση της οδηγίας 2011-36 δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως ε, στις ε, ε πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούνται. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο ε, Δράσης για την καταπολέμηση της ε, λαθρέας διακίνησης μεταναστών ε, αφορά περισσότερο συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, γυναίκες και παιδιά για παράδειγμα, χωρίς όμως να λαμβάνει υπέψη τις διαρθρωτικές συνθήκες που οδηγούν στον ευάλωτο χαρακτήρα της ε, κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο κάθε μετανάστης. Επίσης, ε, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική περιλαμβάνει πολύ σημαντικά στοιχεία, δεν περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την ε, προστασία των θυμάτων και την απροϋπόθετη αρρωγή. Στη, στη μελέτη μας λοιπόν διαπιστώνουμε ότι η το Ευρωπαϊκό Θεματιλόγιο για τη Μετανάστευση και την Ασφάλεια το τράφικινγκ ε, αντιμετωπίζεται ως ε, μορφή οργανωμένου εγκλήματος αλλά δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ε, θυμάτων και των ενδυνάμει θυμάτων. Επίσης, η ευρωπαϊκή αυτή ατζέντα αντιμετωπίζει τα ριζικά αίτια αυτής της μετανάστευσης ε, μέσω της ε, φύλαξης των ε, συνόρων και της καταπολέμησης των διακινητών. Ενώ είναι σαφές ότι το κλείσιμο των συνόρων ενισχύει παρά προλαμβάνει τη λαθρέα διακίνηση ανθρώπων και δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν ασφαλείς διάδρομοι πρόσβασης στην Ευρώπη για αυτούς τους μετανάστες. Τέλος, τονίζουμε πως οι ευρωπαϊκές πολιτικές για το άσυλο ε, ενισχύουν πολλές φορές τον ευάλωτο χαρακτήρα των μεταναστών για εκμετάλλευση, ιδίω στον ε, γεωργικό τομέα. Ε, η, η, χαμηλή ρυθμή λοιπόν επαναπατρισμού δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση μέσω των hot spot πρέπει να αναθεωρηθεί και να δοθεί περισσότερη ε, βάση στην, ε, στην αρχή της ε, ασφαλούς χώρας καταγωγής προκειμένου να μπορούν περισσότεροι μετανάστες να έχουν πραγματικά πρόσβαση στο σύστημα ασύλου και να μην παραμένουν εγκαταλειμμένοι σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στη μελέτη μας επίσης αφιερώσαμε ένα τμήμα σε κάποιες ενδιαφέρουσες εθνικές πολιτικές, κάποιες καλές πρακτικές σε εθνικό επίπεδο που έχουν ως στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και του τράφικινγκ και την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων. Λόγω του ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, δεν μπορώ να σας τα αναφέρω όλα με λεπτομέρειες, αλλά θέλω να σας αναφέρω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Συγκεκριμένα, επικεντρωθήκαμε στην Ιταλική νομοθεσία που, προβλέπει, που παρέχει στα θύματα βοήθεια με, παραμονή, με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ανεξάρτητα ε, από την, ε, το επίπεδο συνεργασίας τους στις ποινικέ διαδικασίες. Ταυτόχρονα ε, η, η προσέγγιση αυτή υποσκάπτεται λόγω της ανεπαρκούς εφαρμογής αυτής. Μια άλλη σημαντική βέλτιστη πρακτική είναι η, η αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου για την καταπολέμηση της ε, κατάχρησης στον χώρο εργασίας που ε, ρυθμίζει τις δραστηριότητες των παρόχων ε, εργατικού δυναμικού μέσω ενός συστήματος αδειοδότησης που έχει ως στόχο την πρόληψη της εκμετάλλευσης. Επίσης, ιδίως στο ιταλικό πλαίσιο αναδεικνύουμε στη μελέτη μας ε, κάποιες πρακτικές που εφαρμόζουν τοπικές ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών για την προστασία των ε, μεταναστών, των εργαζομένων. Λόγω περιορισμού δεν μπορώ να σας τα πω όλα, αλλά θέλω να αναδείξω την πολύ σημαντική δράση της Ομοσπονδίας Πρόξιμα στην Ραγκούζα που μάλιστα ανέπτυξε και μια υπηρεσία μεταφορών για μετανάστριες που εργάζονται στα θερμοκήπια και μάλιστα ε, δημιούργησε και ένα σύστημα με σχολικά λεωφορεία για τα παιδιά που ζουν με τις οικογένειές τους στις περιοχές αυτές. Συμπερασματικά λοιπόν, στη βάση των ε, πορισμάτων της μελέτης μας ε, ολοκληρώσαμε τη μελέτη μας τονίζοντας ότι ο μόνος τρόπος για να προλάβει κανείς και να αντιμετωπίσει την εκμετάλλευση στον γεωρικό τομέα είναι η εφαρμογή μιας πλειάδας ε, δράσεων όχι μόνο δηλαδή η ποινική δίωξη των παραβάσεων αλλά μια, ένα σύνολο δράσεων το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του τη διάσταση του φύλου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και που θα αντιμετωπίζει τους διαρθρωτικούς, τους δομικούς παράγοντες που καταλήγουν στην εκμετάλλευση και στην κατάχρηση ε, που υφίστανται αυτές οι γυναίκες. Και έτσι καταλήξαμε και σε κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις προς τα ε, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν μπορούμε να σας τα παρουσιάσουμε όλα με λεπτομέρειες, αλλά στη διάρκεια της συζήτησης, αν έχετε και εσείς απορία, είμαστε στη διάθεσή σας για να σας τα παρουσιάσουμε. Ευχαριστώ πολύ και τις δύο μιλήτρες για την παρουσίαση της μελέτης. Και ε, τώρα ε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, πολύ λίγο. Ε, θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, να γίνει μια σύντομη συζήτηση και να απαντήσετε στη συνέχεια. Δύο λεπτά, κάστη. Κυρία Κομισάρη, πρώτη, σε σχέση με το ερώτημα που μου απευθύνατε πριν από λίγο για τις διαφορές στο μισθό μεταξύ ανδρών και γυναικών, πέρα από κάποιες συγκεκριμένε περιπτώσεις, ειδικά για τις γυναίκες από τη Ρουμανία, που όπως σας είπα πλέον είναι η πλειοψηφία στην Ραγκούσα, οι γυναίκες αυτές σαφώς πληρώνονται λιγότερο από τους άντρες. Αυτό είναι σαφές. Και αυτό όμως επειδή υπάρχουν και όλοι αυτοί οι διαμεσολαβητές, οι οποίοι πέρα από τα διαβατήρια και τις ταυτότητές τους, κρατάει και μέρος του μισθού τους. Εγώ είχα τη δυνατότητα να δω ότι, ε, και αυτό είναι περίεργο, πολύ συχνά έχουμε συμβάσεις, ειδικά για τις γυναίκες από τη Ρουμανία, επειδή όμως καταφέρνουν να τις εκμεταλλευτούν ακόμα περισσότερο μέσω συμβάσεων τελικά μία από τις γυναίκες η οποία αποφάσισε να καταγγείλει την εργοδότη της ήταν από αυτές που είχαν ε, ένα κανονικ... μια κανονική σύμβαση, 30 ευρώ την ημέρα αμοιβόταν η γυναίκα αυτή, περισσότερο δηλαδή από τις υπόλοιπες γυναίκες. Η γυναίκα επίση αυτή είχε έξι παιδιά, τα οποία τα είχε αφήσει πίσω στη Ρουμανία. Αλλά ακριβώ επειδή είχε τη σύμβαση αυτή, ο εργοδότη την εκμεταλλευόταν ακόμα περισσότερο. Ακριβώ επειδή είχε και ένα μισθό υψηλότερο από τι άλλε γυναίκε θεωρούσε ότι θα έπρεπε να αποδεχθεί μια κατάσταση εκμετάλλευσης την οποία την είχε υποβάλει ο εργοδότης της. Και όσον αφορά τώρα τις κυρώσεις και τις ποινές, επανέρχομαι στην περίπτωση της γυναίκας αυτής, η οποία μετά από δέκα χρόνια συνεχιζόμενης κακοποίησης και εκβιασμών από τον εργοδότη της και μετά από έξι αμβλώσεις και αποβολές αποφάσισε να καταγγείλει τελικά τον εργοδότη της, ο αρμόδιος δικαστής ζήτησε να επιβληθεί στον εργοδότη μια ποινή η οποία είχε να κάνει με συνθήκες ανθρώπινης δουλείας. Η γυναίκα αυτή ήταν έγκλειστη σε αυτό το θερμοκήπιο. Κάθε βράδυ ερχόταν ο εργοδότης και τη ζητούσε σεξουαλικές χάρες εκεί στο θερμοκήπιο που έμενε όταν αποφάσισε λοιπόν η γυναίκα αυτή να τον καταγγείλει, χάρη σε έναν ιερέα από τη Ρουμανία, ο οποίος ζούσε και αυτός σε αυτή την περιοχή και στην οποία τελικά απευθύνθηκε καταφέρνοντας να συγκεντρώσει όλο το θάρρος που της είχε απομείνει για να καταγγείλει τον εργοδότη της, η ποινή που επελέγει για τον εργοδότη αυτή ήταν μια ποινή η οποία αντιστοιχεί σε ε, συνθήκες καταναγκαστικής ε, δουλείας. Υπάρχει λοιπόν η κατάλληλη νομοθεσία στην ε, Ιταλία, αλλά το πρόβλημα είναι ότι επιβάλλεται μόνο σε περιπτώσεις ε, σεξουαλικής βίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις όταν ε, καταδικάστηκαν τελικά εργοδότες, καταδικάστηκαν για λόγους σεξουαλικής βίας και κακοποίησης και όχι για λόγους αναγκαστικής δουλείας. Η Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βουλευτές. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης που ακούσαμε προηγουμένως, η Βιωρή Κανταντσίλα, πρωθυπουργός της Ρουμανίας, νυν και πρώην Ευρωβουλευτής, ε, ακούσαμε ότι ε, πήγε στη Ρακούζα, ε, σε μια περιοχή όπου τότε εργάζονταν 7.500 Ρουμάνες. Και στη συνέχεια ανέλαβε δράση η, η κυβέρνηση. Υπάρχει μια οργάνωση τοπική που λέγεται Πρόξιμα και για την οποία ακούσαμε προηγουμένως και ασχολείται με την προστασία των ε, Ρουμάνων ε, γυναικών στη Ραγκούζα έχει ε, υπάρξει και ενημερωτική εκστρατεία στην βόρειο-ανατολική Ρουμανία από όπου κατάγονται οι γυναίκες αυτές που πηγαίνουν στη Ραγούζα. Και όπως σας είπα, έχουμε κάνει και ενημερωτική εκστρατεία ευαισθητοποίησης σε όλη τη χώρα. Οι ρουμανικές αρχές, σε συνεργασία με τις Ιταλικές αρχές, προχώρησαν όμως ακόμα περισσότερο με επιτόπιους ελέγχους στις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις όπου προέκυψε η εξής ε, κατάσταση. Οι περισσότερες παράνομα εργαζόμενες μετανάστριες από τη Ρουμανία αρνήθηκαν όχι μόνο να κάνουν μήνυση στην Ιταλική αστυνομία αλλά να συζητήσουν καν για το θέμα. Βλέπετε πόσο ευάλωτες είναι και σε τι καταστάσεις εκτίθενται. Μετά από αυτή την ενημερωτική εκστρατεία λοιπόν στη Ρωμανία και τους επιτόπιους ελέγχους στη Ραγκούζα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η κατάσταση έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Δεν μπορούμε παρά να είμαστε αισιόδοξοι. Θα διατηρήσουμε τα μέτρα που έχουμε ε, λάβει έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των γυναικών αυτών, όχι μόνο στην Ιταλία και αλλού. Σε σχέση με το όσα είπε η κυρία από τη Σουηδία για τα παιδιά και το πόσο ευάλωτα είναι. Έχουμε αρμόδιο φορέα για την προστασία των ανηλίκων στη Ρουμανία ε, που μας έχει κάνει μια έκθεση για την κατάσταση αυτή. 95.000 είναι τα παιδιά από τη Ρουμανία ε, τα οποία αυτή τη στιγμή ε, τα έχουν εγκαταλείψει ουσιαστικά οι γονείς τους στη Ρουμανία ε, για να εργαστούν στο εξωτερικό, νόμιμα ή και παράνομα καμιά φορά. Ακούσαμε ε, για τις κυρώσεις ε, οι οποίες επιβάλλονται στους διαφερούς ενδιαμέσους στα πρακτορία που παρέχουν εργατικό δυναμικό στην Ισπανία και την Ιταλία. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι ίδιες οι εργαζόμενες ε, αντιστέκονται. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά και οι ίδιοι, υπάρχουν κάποιοι ε, διακινητές, κάποιοι εκμεταλλευτές, ε, σύγχρονοι δουλέμποροι ε, που έχουν όλη τη δραστηριότητα. Ακούσαμε την παρουσίαση της μελέτης αμέσως πριν και για τη Ρουμανία, η Ιταλία και η Ισπανία είναι προορισμοί που επιλέγουν οι εργαζόμενοι μας. Αυτή τη στιγμή πραγματικά αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για τη Ρουμανία γιατί δεν βρίσκουμε εργαζομένους. Έχουμε 200.000 θέσεις εργασίας που μένουν ελεύθερες. Αυτά τα λέει ε, το Υπουργείο Εργασίας. 200.000 θέσεις εργασίας στη Ρουμανία δεν βρίσκουν εργαζομένους. Και η Ρουμανία σέβεται το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων όπως αναφέρεται ε, στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στο άρθρο 23. Αυτό αναφέρεται και στο άρθρο 23 του Ρουμανικού Συντάγματος. Ευχαριστώ. Ε, καθηγήτρια κυρία Σολτάρ. όχι πάνω από δύο λεπτά. Έχουμε και άλλο θέμα στην ημερησία διάταξη. Πρέπει να τελειώσουμε αυτό εδώ. Δύο, δύο πολύ σύντομα σχόλια μόνο. Αναφέρθηκα σε μία έρευνα προηγουμένως όπου βρήκαμε διαφορές στις αμοιβέ ε, με βάση το φύλλο, ε, κανονικά αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει γιατί έχουμε διαφορά στους μισθούς στην επίσημη αγορά εργασίας και γιατί να μην υπάρχει αυτό και στην ανεπίσημη, δηλαδή στη μαύρη εργασία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που αναφέρεται στη δική σας έκθεση είναι πραγματικά εξαιρετική η μελέτη από ό,τι ακούω και βλέπω και αυτό που βρήκα ενδιαφέρον είναι ότι μιλάτε για τα νομικά εργαλεία και πώς είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν ε, τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών και των ετούντων άσυλο που καταφθάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ότι είναι καλύτερη προστασία προς τους ανθρώπους αυτούς από ότι για τους ίδιους τους Ευρωπαίους εργαζομένους και μάλιστα τις γυναίκες που εργάζονται στη Γεωργία. Είναι νόμιμες μετανάστριες είναι εργαζόμενες που κυκλοφορούν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που τις προστατεύουμε χειρότερα από ότι τους παράτυπους, ας πούμε, μετανάστες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλες τις ομιλήτριες για τις παρουσιάσεις και ε, τη μελέτη, πολύ ενδιαφέρουσα. Στόχος της παρούσας ακρόασης ήταν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης αυτών των γυναικών. Πώς να προστατεύονται καλύτερα ε, και πώς να ενημερώνονται. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή, πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο. Και στα κράτη-μέλη. Και οι εθνικές αρχές έχουν ευθύνη και οι τοπικές αρχές ε, όλοι πρέπει να συνεργάζονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Επόμενο θέμα μερίσια διάταξη. Μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη ηθική και τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασία, σε δημόσιου χώρου και στην πολιτική ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξέταση του σχεδίου έκθεση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μα, την κυρία Πίνα Πιτσιέρνο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω σύντομα να σε εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους θελήσαμε τόσο πολύ να συντάξουμε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεώρησα καταρχά ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί η φωνή των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίω της δικής μας της Επιτροπής μια φωνή που θα έπρεπε να υποστηρίξει τα εκατομμύρια των γυναικών που συντάχθηκαν με το κίνημα MeToo, το κίνημα αυτό καταγγελίας για την ηθική και σεξουαλική παρανόχληση. Θεώρησα όμως ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να αντιταχθούμε και στον ε, μοραλισμό αυτό που ε, προέβαλαν διάφοροι άλλοι αν θέλετε παράγοντες οι οποίοι συνεχίζουν και λένε ότι μα οι γυναίκες πήγαιναν γυρεύοντας. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει για άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι οι γυναίκες είναι δύο φορές θύματα. Θύματα τη στιγμή που δέχονται την κακοποίηση και την παρενόχληση, αλλά θύματα μια δεύτερη φορά όταν ε, καταδικάζονται βασικά και επικρίνονται για αυτά τα οποία λένε, για αυτά τα οποία φοράνε, για τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζουν επειδή δεν είχαν τη δύναμη να κάνουν μια καταγγελία τη στιγμή της παρενόχλησης. Οι γυναίκες αυτές, κυρίες και κύριοι, ουσιαστικά είναι μία από εμά. Μπορεί να είναι διάσημες ή άγνωστες, μπορεί να είναι πλούσιες ή φτωχές, μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε οικονομική ή κοινωνική τάξη, από οποιοδήποτε φίλη, από οποιοδήποτε μορφωτικό υπόβαθρο. Από πουδήποτε και αν προέρχονται οι γυναίκες αυτές, όλο και περισσότερο αποτελούν θύμα παρενόχλησης, ηθικής, σεξουαλικής, έμεσης, άμεσης, οι γυναίκες αυτές αναγκάζονται να αποδεχθούν συνθήκες απαράδεκτες για την ελευθερία τους, για την σταδιοδρομία τους, συνθήκες απαράδεκτες για την ίδια τη ζωή τους. Αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά μία πολύπλοκη πρόκληση γιατί τα αριθμητικά δεδομένα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καταδεικνύουν πραγματικά ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Όλες οι έρευνες που έχουν γίνει στον τομέα αυτό μας λένε ότι μία στις δύο γυναίκες στην Ευρώπη έχουν ήδη πέσει θύμα παρενόχληση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στρατηγικές όχι μόνο καταπολέμησης αλλά και πρόληψη του φαινομένου. Και αυτό διότι η μορφή που παίρνουν όλες αυτές οι παρενοχλήσεις αλλάζει συνεχώς με την πάρδα του χρόνου. Εξελίσσεται η παρενόχληση τελικά και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν και αυτές με τη σειρά τους στην αύξηση των φαινομένων ηθικής παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης. Ας μην ξεχνάμε όλες αυτές τις περιπτώσεις καταγγελιών μέσω του Twitter, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά τα φαινόμενα του ε, εκδικητικού πορνό που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν πάρα πολλοί που χρησιμοποιούν πλέον όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες. Υπάρχουν νέες μορφές λοιπόν παρενόχλησης που ε, θα πρέπει να καλυφθούν από νέες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να προσαρμοστούν δηλαδή οι στρατηγικές μας. Ας μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκε αυτή τη στιγμή δέχονται παρενόχληση όχι μόνο στο χώρο εργασία, αλλά και στο δρόμο, στα μπαρ, στα εστιατόρια, σε όλε τις εκφάνσει τη ε, δημόσια και ιδιωτική του ε, ζωή σε ορισμένες περιοχές του κόσμου δεν προβλέπονται συγκεκριμένες στρατηγικές. Σε άλλες ε, χώρες δειλά-δειλά αρχίζουν σιγά-σιγά να εμφανίζονται κάποιες στρατηγικές προστασίας των γυναικών. Βλέπουμε όμως ότι ένα κίνημα έχει ήδη ξεκινήσει. Ο εκφοβισμός, η παρενόχληση, η ηθική και σεξουαλική βασίζεται βασικά σε φαινόμενα διακριτικής μεταχείρισης, σε μια διαφορετική αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών, σε μια εγγενή διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών. Επομένως, δεν θα πρέπει να βλέπουμε τις ε, εκδηλώσεις αυτές, την παρενόχληση αυτή, μόνο την ύπαρξη μιας πατριαρχικής κοινωνίας, αλλά και το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει αρκετά η χειραφέτηση των γυναικών. Προφανώς πάρα πολλά πράγματα έχουν γίνει και στο Κοινοβούλιο και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη για να καταπολεμήσουμε το στίγμα που βαρύνει πάρα πολλές γυναίκες, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ακόμα ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις παρενόχλησης και εκφοβισμού στο χώρο εργασίας που δεν καταφέρνουμε να εξαλείψουμε και που δεν καταφέρνουμε να καταδικάσουμε. Αναφερθήκαν πριν από λίγο σε, όλες αυτά τα, όλα αυτά τα φαινόμενα που έχουμε στο γεωργικό τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταδικάσουμε τις παρενοχλήσεις αυτές, γιατί αν δεν το κάνουμε, ουσιαστικά υπονομεύουμε και υποσκάπτουμε μία ακόμη φορά τη θέση των γυναικών. Είναι ουσιαστικά σαν να μην αποδεχόμαστε ότι είναι ίσοι άνδρες και γυναίκες. Ο σεξισμός και η παρενόχληση θα πρέπει καταρχάς να αντιμετωπιστούν κυρίως σε επίπεδο πολιτισμικό, σε επίπεδο νοτροπίας. Θα πρέπει να καταρρύψουμε όλα αυτά τα εσφαλμένα, παροχημένα στερεότυπα κατά των γυναικών. Και κάτι ακόμα το οποίο το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα κουραστώ ποτέ να το λέω, αν ακόμα και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν ακόμα και στα πλαίσια της Ολομέλειας, πολλές φορές ακούμε ρητορική, σεξιστική από άνδρες συναδέλφους, αυτό από μόνο του τελικά τι σημαίνει, ότι μας περιμένει τεράστια εργασία ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια εργασία πολύ μεγάλη, μια εργασία πάρα πολύ δύσκολη, την οποία όμως πρέπει να κάνουμε. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολιτισμική τελικά η προέλευση των διακρίσεων που έχουμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και που μπορεί να οδηγήσει σε εκφοβισμό, μπορεί να οδηγήσει σε παρενόχληση, μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορές επιβλαβής για τις γυναίκες στο δημόσιο και ιδιωτικό τους βίο. Καταλαβαίνετε το σημαντικότατο ρόλο που διαδραματίζει η παιδεία και είναι πάρα πολύ σημαντικό από τους παιδικούς σταθμούς μέχρι το πανεπιστήμιο, μέχρι τα προγράμματα κατάρτισης που έχουμε στον χώρο εργασίας να ενσωματώνει τη διάσταση αυτή υπεράσπισης ε, των γυναικών. Οι περισσότερες γυναίκες γνωρίζουν ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το να βρούμε έναν κοινό νομικό ορισμό όσον αφορά την παρενόχληση. Ένα νομικό ορισμό για όλα αυτά τα φαινόμενα γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έναν κοινό ορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίος θα μας επέτρεπε να συγκρίνουμε κάπως το φαινόμενο αυτό από τη μία χώρα στην άλλη. Χάρη στο κίνημα MeToo βλέπουμε ότι από κοινωνική τουλάχιστον πλευράς υπάρχει μια νέα συνειδητοποίηση του τι σημαίνει να είναι κανείς θύμα παρενόχλησης. Δυστυχώς η συνειδητοποίηση αυτή δεν υπάρχει ακόμα σε νομικό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρξει και εκεί. Εγώ αυτό προσπάθησα να τονίσω στο σχέδιο έκθεση το οποίο έχετε ενώπιόν σα και πιστεύω και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι σημαίνει δημόσιο χώρο. Τι στη δημόσιο χώρο. Αυτή τη στιγμή πέρα από του κλασικού δημόσιου χώρου έχουμε και του εικονικού δημόσιου χώρου στο διαδίκτυο όπου οι γυναίκε όλο και περισσότερο υφίστανται παρενόχληση. Αναφέρθηκα, αναφέρθηκα στο τι γίνεται σε πάρα πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό λοιπόν το τονίζω στα πλαίσια της έκθεσής μου. Ελπίζω ότι με τις δικές σας τις τροπολογίες θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε περισσότερο το, το κείμενο αυτό το οποίο έχω υποβάλει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχουν οι σκιώδεις Η κυρία Ζαμπόρσκα είναι η σκιώδης από το ΕΛΚΑ. Ε, την εκπροσωπεί όμως ε, η κυρία... E, ε, Ζαμπόσκα δεν μπόρεσε να έρθει ε, σήμερα για να σας παρουσιάσει την απόψη της. Θα τα παρουσιάσω εγώ. Χαιρετίζει το έργο της εισηγήτριας, η κυρία Ζαμπόσκα, και τις προσπάθειες που κατέβαλε για να ε, συντάξει αυτή την έκθεση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως παρουσιάζει τα αρνητικά και τα δεινά που υφίστανται οι γυναίκες, αλλά από την άλλη προτείνει ή τουλάχιστον αναζητεί ε, τις ενδεχόμενες λύσεις. Η κυρία Ζαμπόσκα λυσεις ότι ε, παίζουν κομβικό ρόλο οι άνδρες στην ε, αναζήτηση των λύσεων και στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ενημερωτικέ εκστρατείε προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης η κυρία Ζαμπόρσκα θεωρεί ότι Υπάρχουν πολλοί τρόποι καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Υπάρχει και η ψυχολογική βία, το mobbing ε, και η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Πάντως υπάρχει ένας ευρύτερος στόχος, ε, η εξάλληψη κάθε είδους βίας κατά των γυναικών και άλλων ευάλωτων μελών της κοινωνίας. Η κυρία Ζαμπόρσκα έχει κάποια σχόλια και κάποιες ε, ανησυχίες ε, για την ορολογία για την επικουρικότητα και θα τις καταθέσει προσεχώς. Η κυρία Μπεσέρα από την ε, ομάδα των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Πιτσέρνο. Είναι πραγματικά εξαιρετική η εργασία της εδώ. Εγώ ήμουν σκιώδης εισηγήτρια των Φιλελευθέρων για την καταπολέμηση ε, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και παρενόχλησης τον Οκτώβριο για το αντίστοιχο ψήφισμα και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία τώρα να συνεργαστώ με την εισηγήτρια. Ξέρουμε ότι ο εκφοβισμός και η παρενόχληση ε, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και στους χώρους εργασίας αλλά και στη δημόσια ζωή γενικότερα. Έχουν γίνει πολλές πρόοδοι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 30 έτη, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να κατανοήσουμε τι ακριβώς γίνεται. Ε, όταν πρόκειται για τέτοιο εκφοβισμό και σεξουαλική παρενόχληση, υπάρχει ένα μοντέλο αντίδρασης που είναι η σιωπή, ε, η ε, συνενοχή και η ενοχοποίηση των θυμάτων. Επίσης υπάρχει ε, μια άνηση ε, θέση των γυναικών ε, στις διάφορες σχέσεις εξουσίας. Πολλές φορές τα θύματα ή και οι ίδιοι μάρτυρες διστάζουν να καταθέσουν γιατί φοβούνται να μην χάσουν τη δουλειά τους. Ε, και πολλές φορές η κοινωνία σκέφτεται, δικάζει, κρίνει και καταδικάζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεν ισχυρή νομοθεσία, αλλά δυστυχώς τα κράτη-μέλη δεν την εφαρμόζουν πάντα ε, με συνέπεια ως όφιλ. Στηρίζουμε αυτό που ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, η συγγήτρια, να βελτιωθούν οι μηχανισμοί ελέγχου, έτσι ώστε να εφαρμόζεται σωστά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που απαγορεύει τη σεξουαλική παρενόχληση. Όπως είδαμε πρόσφατα σε μια υπόθεση στην Ισπανία, θα πρέπει κατεπηγόντως ε, ε, να έχουν κοινού ορισμούς τα κράτη-μέλη. Και σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τη συνένεση και για τους άλλους ε, ορισμούς. Επίσης ανησυχώ πολύ ε, ε, για την παρενόχληση στα κοινωνικά δίκτυα και στον κυβερνοχώρο, γιατί αφορά ε, ιδιαίτερα και με δυσανάλογο τρόπο τις γυναίκες και τα κορίτσια. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν πολιτικές πρόληψεις που να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και αυτό είναι υποχρέωση από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η ομάδα μας ε, καλεί μετεπιτάσεως τα κράτη-μέλη που ακόμα δεν έχουν συμβασ... Ε, κυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης να το πράξουν και να μην μπλοκάρουν στο Συμβούλιο τη σχετική απόφαση. Επίσης, θα πρέπει να διευρυνθεί ο ορισμός ε, της ρητορικής μίσους, που είναι και παράνομος είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες αυτή της Επιτροπής Γυναικών για, ε, για το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2019. Άλλη προτεραιότητα να προταθεί μια οδηγία κατά κάθε είδους ε, βίας κατά γυναικών και κοριτσιών και η έμφυλη βία. Αυτά όλα είναι στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα ζητάμε, έχει έρθει η ώρα επιτέλους να γίνουν. Ε, θέλουμε να πιέσουμε προς όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου για να εφαρμοστεί ε, το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου και ε, μέχρι τώρα η πρόοδος ήταν υπερβολικά αργή, ανεπαρκής και όλα αυτά είναι απλούστατα απαράδεκτα. Στο Κοινοβούλιο ιδιαίτερα. Είναι στόχος να προστατεύσουμε, να βοηθήσουμε τα θύματα και να ε, προωθήσουμε τη μηδενική ανοχή. Να σπάσει η σιωπή. Με, το κίνημα MeToo έχει ανοίξει μια χαραμάδα σε αυτό το τοίχο αλλά θα πρέπει εμείς κάθε μέρα να βάζουμε μια σφήνα για να διευρύνεται αυτό το ε, ε, ρήγμα και το άνοιγμα για να προστατευτούν επιτέλους τα θύματα. Τέλος θέλω να θυμίσω ότι ε, περιμένω στις 20 Ιουνίου την σχετική ακρόαση. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Σολέ από τους Πρασίνους. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή ε, αφορά ένα πολύ σημαντικό, τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, πρόβλημα μεγαλύτερο από ό,τι μπορεί κανείς να ε, υποψιαστεί με μια πρώτη ματιά. Γενικά, τα, τα, οι υποθέσεις ε, σεξουαλικής παρενόχλησης που έχουν έρθει στην ε, επιφάνεια ε, είναι πάρα πολλές από το Hollywood μέχρι την Ισπανία. Ε, αυτές οι υποθέσεις έχουν λάβει μεγάλη δημοσιότητα μέσα των μέσων ενημέρωσης, πολλές αντιδράσεις, αλλά να μην ξεχνάμε ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων, των υποθέσεων αυτών δεν αποκαλύπτονται ποτέ και ε, παραμένουν κρυμμένες. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου στα χαρτιά έχουμε επιτύχει κάποιες σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Δυστυχώς όμως η ίδια η δομή της κοινωνίας μας εξακολουθεί να βασίζεται σε πατριαρχικές ε, δομές που εμποδίζουν την πλήρη ισότητα. Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί ε, μια κατάφορη εκμετάλλευση ε, δομών εξουσίας που πρέπει να αναδιαμορφωθούν και να αλλάξουν και πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε ε, αυτή την κουλτούρα βίας που υπάρχει στην κοινωνία μας. Ε, ως ε, σκιώδη λοιπόν εισηγητή εκ μέρου των Πρασίνων θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την παρουσίαση της έκθεση, την χαιρετίζω. Νομίζω ότι είναι μια ολοκληρωμένη έκθεση που θα αποτελέσει καλή βάση για τις από εδώ και πέρα εργασίες μας και θέλω να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλούμε ανοιχτά για την ε, σεξουαλική παρενόχληση και βία στην πολιτική ζωή και στους πολιτικούς θεσμούς δηλαδή γιατί ξέρουμε ότι συμβαίνουν τέτοια περιστατικά και εκεί και εμείς ως ερετοί εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών λαών έχουμε καθήκον να, καταπολεμήσουμε αυτές ε, αυτά τα περιστατικά. Με τις τροπολογίες μας θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έμφαση σε κάποια συγκεκριμένα θέματα, για παράδειγμα εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ε, εκπαίδευσης, όχι μόνο για δικαστές και αξιωματούχους επιβολής του νόμου, αλλά και για ε, στελέχη των πολιτικών κομμάτων. Ε, σχέδια δράσης και πρόληψης εντός των πολιτικών θεσμών και των πολιτικών κομμάτων, ε, επαρκείς διαδικασίες και εχέγγυα για, για να μπορεί μια γυναίκα να καταγγείλει αν της συμβεί κάτι τέτοιο, ε, σοβαρή στήριξη των θυμάτων και ανάγκη ύπαρξης ενός ισχυρού νομοθετικού πλαισίου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε αυτά τα θέματα λοιπόν θα εστιάσουμε εμείς την προσοχή μας ε, μέσα από τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος στην εισηγήτρια. Δύο με τρία λεπτά, όχι παραπάνω όμως. Σας παρακαλώ.